Dear colleagues, it is uh, time to start. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Με αυτό ξεκινάμε είναι κάτι που το αναμένουν διακαώς πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Σημείο 13 στην εμείς διάταξη, προφορική ερώτηση για τις πάνιες μορφές ανταλλαγή μάλλον απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο κανονισμού τη Επιτροπή τροποποιεί τον κανονισμό αριθμό 692-2008 σχετικά με τι εκπομπέ από ελαφρά επιβατικά και εμπορικά οχήματα Euro 6 όπω είναι γνωστό. Το έχουμε συζητήσει αυτό το σημείο σε προηγούμενες συνεδριάσεις για το πραγματικό ζητούμενο είναι η διαδικασία για τις ε, εκπομπές σε συνθήκες οδήγησης, τι ε, τις πραγματικές δηλαδή εκπομπές. Και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια σχετική δέσμη μέτρων κατά τη διάρκεια του 2016. Έχουμε όμως ακούσει κάποιες πληροφορίες για τη διαδικασία των πραγματικών συνθηκών οδήγησης και πώς υπολογίζονται σχετικά οι εκπομπές, τους ε, φορείς, τους παράγοντες ε, συμμόρφωσης που θα θέλαμε να μας τους εξηγήσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα νομίζω μπορούμε να δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας εξηγήσει τη νέα της πρόταση. Αργότερα θα συζητήσουμε με τα μέλη της Επιτροπής και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και ερωτήσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω θα το περιμένατε. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Ο κύριος Κοζίκου, Διευθυντής, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 28 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Μηχανοκίνητων Οχημάτων είναι ένα παράδειγμα που δείχνει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα περιβάλλον, ένα σκηνικό αρκετά ε, δυσχερές. Η ψηφοφορία είναι το πέρας ε, μιας δουλειάς που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια για το νέο κείμενο, στα πλαίσια της εντολής που έχει απονατεθεί από τους συνομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό Euro 6, το κείμενο για τις εκπομπές σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης, RDE, τα αρχικά. Για το οξύδιο του αζότου, NOx, τα όρια έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά από το 2010, διότι από το 2010 στο 2014 οι προδιαγραφές ε, γύρω 3 ε, και 6 προέβλεψαν όρια που πέρασαν από 500 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο σε 400 ε, μιλιγκράμμ. Για τα οχήματα που κινούνται με δίζελ όμως έχουμε τετραπλάσιες τιμές από αυτές που είναι οι οριακές αυτή τη στιγμή όταν μετρούμε ε, το τι γίνεται σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης από τι εργαστηριακές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να θεωρήσουμε τις δοκιμές για να αντικατοπτρίζεται ο όγκος των εκπομπών σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης εξού και τα τεστ RDE. Η διαδικασία αυτή θα συμπληρώσει τις εργαστηριακές δοκιμές και θα επιτρέπει σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης να δούμε τα επίπεδα των εκπομπών οξυδίων του αζότου σε ένα μεταγενέστερο μάλιστα στάδιο και τον αριθμό σωματιδίων. Οι δοκιμές πραγματικής οδήγησης θα επιτρέψουν να μειωθούν αισθητά οι σημερινές παρεκκλήσεις καθώς και ο κίνδυνος παραποίησης των συστημάτων που ισχύουν. Ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί πρόσφατα με τις διάφορες ε, συσκευές που ε, μετρούν τις εκπομπές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη γεωγραφική περιοχή ε, στον κόσμο που προβλέπει τόσο αυστηρές δοκιμές. Η νέα διαδικασία ε, ψηφίστηκε τον Μάιο 2015 από την Επιτροπή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και θα αρχίσει να ισχύει από το 2016, τον Μάιο. Ε, δεν θα έχει ακόμα αντίκτυπο για την κατασκευή οχημάτων, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για να τελειοποιήσουμε στην πράξη τις γνώσεις μας μετά από τους ελέγχους και τις δοκιμές. Οι φάσεις της πραγματική υλοποίησης θα έχουν ομοτατικές συνέπειες καθώς και στα μέγιστα όρια των εκπομπών και αυτά ορίστηκαν όπως σας είπα στις 28 Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία αυτή είναι η βάση επί της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην ε, οργάνωση των ελέγχων μετά από την εξέταση βεβαίως της πρότασης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2007 είχαν προβλεφθεί νέες ε, από το 2017 μάλλον θα προβλεφθούν ε, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των δοκιμών για την εμπορία και την κατασκευή των νέων οχημάτων και το 2019 για όλο ε, το στόλο οχημάτων. Από το 2017 έως 2019 θα είμαστε στα 110%, 50% για τα νέα μοντέλα ε, το 2019 και από το 2021 για όλα τα οχήματα. Θα υπάρχει βεβαίω και μια μεταβατική περίοδο για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκέ αυτοκινητοβιομηχανίε να προσαρμοστούν επαρκώ και να λάβουν υπόψη τα τεχνικά όρια για τι ε, πραγματικέ ε, εκπομπέ των οχημάτων που κινούνται με δίζελ. Περιμένουμε και σημαντικότερες μειώσεις, αλλά χρειάστηκε να βρεθούμε και κάποιου συμβεβασμού για να υπάρξει γρήγορη επίλυση του θέματος και να προβλέψουμε σύντομα αυστηρούς έλεγχους που είναι οι προτεραιότητα, προτεραιότητές μας. Αν δεν υπήρχε συμφωνία θα ίσχυαν οι σημερινοί κανόνες και οι σημερινοί έλεγχοι. Η συμβαστική λοιπόν λύση θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση των εκπομπών οξυδίων του αζότου χωρίς να αλλάξει ο προγραμματισμός παραγωγής μοντέλων από τους αυτοκινητοπαραγωγούς. Χωρίς αυτή τη συμφωνία τα οχήματα diesel θα συνέχιζαν να εκπέμπουν μέχρι 400 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο. Στην πράξη κάτι που συμβαίνει τώρα. Ε, έτσι ε, όλα τα οχήματα θα καλύπτονται από το 2019 στο όριο των 80 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο και λαμβάνοντας υπόψη ε, τους παράγοντες συμμόρφωσης, 168 ε, μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο το 2019, αντί για 400 ε, μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο, δηλαδή 80% σε σχέση με το τι θα ίσχυε χωρίς τα, τους παράγοντες συμμόρφωσης και 120% ε, για το 2021. 120 μάλλον μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο. Επίσης για τις φορητές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές. Εφόσον οι τεχνολογικές λύσεις βελτιωθούν όπως ελπίζουμε, το περιθώριο σφάλματος 50% που αυτή τη στιγμή προβλέπεται θα μειωθεί. Η ετήσια αξιολόγηση προβλέπεται από το σύστημα των ελέγχων και με συμφωνίε των κρατών μελών, ε, τα οποία ενέκριναν τα κάτι μέλη στι 28 Σεπτεμβρίου, στην, ε, Οκτωβρίου μάλλον, στην Επιτροπή των Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη κάποια μέλη έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μία ε, μάλλον με δύο δικές μου τεχνικές ερωτήσεις. Καταρχήν, πότε θα μας κοινοποιήσετε επισήμως στο κείμενο και δεύτερον, θέλουμε λιγότερη τεχνολογία, περισσότερη πολιτική στο κείμενο αυτό. Ξέρετε πως σε κάθε επιτροπή προετοιμάζεται και μία γνωμοδότηση. Πείτε μου λοιπόν για τα οχήματα ε, συμβαίνει αυτό, μπορούμε ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας παρουσιάσατε να την τροποποιήσουμε εκεί. Τι συμβαίνει δηλαδή με αυτή την Επιτροπή Μηχανοκίνητων Οχημάτων, πώς λειτουργεί. Η κυρία Φλόρεντς έχει το λόγο. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα μεγάλη προσοχή την Επιτροπή και πιστεύω κι εγώ ότι ήταν πολιτική η απόφαση. Όσο και να έλειψαν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να εκφράσω την επιθυμία για πιο αυστηρές τιμές στις χρήσεις αυτές που έχει προτείνει η Επιτροπή Ο υπολογισμό φαίνεται ότι είναι καταστροφικό αυτή τη στιγμή και θα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν βλέπει να υπάρχει δυνατότητα να είναι πιο διαφανή συνθήκε διαμόρφωση τιμολόγηση ή αν είναι περίπλοκες οι διαδικασίε όπω με το διεξίδιο του άνθρωπου. Μια απλή ερώτηση πιστεύω μπορώ να περιμένω να λάβω και απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γκρότα. Ευχαριστώ. Θα έχουμε συζητήσει πιστεύω αυτά τα οποία μας ε, προτείνει η Επιτροπή. Είχαμε ένα περιθώριο σε σχέση με την ε, μια ανοχή σε σχέση με την ε, υπέρβαση των ορίων. Τώρα είχαμε το παράγοντα 2,1 για τα οξύδια του αζότου που είχαμε ορίσει το 2006 Τώρα φαίνεται ότι φτάνουμε στο επίπεδο Ευρώπης 5, Γιουρ 5 αντί για 6. Πάμε πίσω δηλαδή σε σχέση με το Γιουρ 6. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να το δεχθούμε αυτό. Δεν μπορεί να παραμερίζεται και να υποβαθμίζεται σε επίπεδο Γιουρ 5 η νομοθεσία μας. Για τα οξύδια του Αζώτου συγκεκριμένα έχουμε την αρμοδιότητα ή καλύτερα την υπευθυνότητα, την ευθύνη του, της ζώνης του όζοντος και την τελευταία εβδομάδα στην Ολομέλεια συζητήσαμε πολλά ζητήματα σχετικά, αλλά οι οριακές τιμές, οριακές τιμές που έχουν ηλικία 10 ετών, τι νόημα έχει να τις συζητάμε και μάλιστα να συζητάμε να τις υποβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τι θέλετε να σε αυτές τις παράνομες ε, επιλογές, για να μην μιλήσουμε για τις παράνομε πρακτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Ξέρουμε ότι όχι μόνο στα οξύδια του αζότου, αλλά και στα όρια στις θέροντες τιμέ ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και ο κύριος ε, Σακώνη, όπω και εγώ είχαμε ασχοληθεί με την αναθέωση του 2013. Τι είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση με τι ωριακέ τιμέ και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοφύλακα των συνθήκων. Τι εργαλεία έχει στη μέση τη. Χρειάζεται να γίνει και άλλη συζήτηση, ευρύτερη συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να δούμε ότι δεν τηρούνται η νομοθεσία, οι τιμέ, αυτά τα οποία είναι χάρτου καταγεγραμμένα και ότι δεν είστε σε θέση να τα ελέγξετε, να επιβεβαιώσετε ότι τηρούνται ή ότι είναι σε θέση τα κράτη-μέλη να βγαίνουν ξαφνικά από μια γωνιά για να πούνε 2,1 ενώ κανείς δεν ξέρει πώς έχει καταρτιστεί αυτό το νούμερο, τι συμπεριλαμβάνει. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αυτή τη συζήτηση και στην Ολομέλεια. Υποτίθεται κάναμε συζήτηση με βάση πραγματικά δεδομένα, με γνώση της υπόθεσης, με, με πραγματογνωμοσύνες και τώρα βλέπουμε μια αδιαφανή διαδικασία προτάσεις αυθαίρετες, οι, οποία, οι οποίες για μας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σημαίνουν ότι πρέπει να πατήσουμε το φρένο αμέσω. Να σταματήσει η διαδικασία, αλλιώς γελιοποιούμεθα. Λοιπόν, για να, για να διατηρηθεί η νομιμότητα και να διατηρηθεί η διαδικασία πρέπει να αποσυρθούν όλα αυτά και να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Ε, έχουμε πλέον την προϋπόθεση για τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, το Real Drive Emission. Έχουμε τα, τις προϋποθέσεις, γιατί 3 Σεπτεμβρίου συζητήσαμε και το είπα, και πάλι στις 24 Σεπτεμβρίου, ότι δεν υπάρχει πεδίο απάτης μεγαλύτερο από αυτό των δοκιμών και παληθεύσεων εκπομπών στο αυτοκίνητο. Χωρίς να έχουν βγει όλα αυτά που βγήκαν μετά στη φόρα. Δεν είναι δυνατόν όμως τώρα να συνεχίσουμε έτσι. Θα πρέπει να δώσουμε ε, μία εξήγηση γιατί δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων που βρίσκονται υπόλογοι για τη μη των προδιαγραφών και για την διαρκή υποβάθμιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και τους δήμους και ότι έχει ανανεωθεί υποτίθεται και ανανεώνεται διαρκώς ο στόλος των ε, οχημάτων με κινητήρα. Γιατί λοιπόν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διαφορές. Και τώρα μας λέτε ότι θέλετε να το επιβεώσετε, να το επικυρώσετε καλύτερα με ένα de facto 2,1 χωρίς καμιά εξήγηση. Νομίζω ότι είναι γελία η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννη, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω τα εξής. Όταν είδα ποια ήταν τα αποτελέσματα της τεχνικής συνάντησης για πρώτη φορά, είχα την εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απογοητευτεί πάρα πολύ από το αποτέλεσμα αυτό. Πάρα πολύ. Γιατί είχαμε ακούσει διάφορες φήμες για την αρχική πρόταση που είχε βάλει στο τραπέζι η Κομισιόν και η τελική μορφή της δεν ήταν καθόλου κοντά στην αρχική πρόταση. Και γι' αυτό με ιδιαίτερη έκπληξη διάβασα το ανακοινωθέν τύπου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου πρώτα απ' όλα ανακοινώθηκε πως είμαστε η πρώτη και η μοναδική περιφέρεια στον κόσμο όπου θα ισχύσουν αυτές οι δοκιμές για τις πραγματικές εκπομπές. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο σεμνοί δεδομένου πως ήταν οι ΙΠΑ οι οποίες μας υπέδειξαν το πρόβλημα και μετά είδα να υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια την απόφαση αυτή η Κομισιόν παρόλο που θεωρούσα ότι θα έπρεπε να έχουν απογοητευτεί τρομερά. Γιατί λοιπόν δεν μπορείτε να ε, ε, καταγγείλετε τα κράτη-μέλη ε, ανοιχτά για το γεγονός πως παίζουν πολιτικά παιχνίδια, πως δεν πέρασε η αρχική σας ε, πρόταση και πως οι παραγόντες συμμόρφωσης ακολουθεί τη δική τους πολιτική λογική και όχι τις επιταγές της Τεχνικής Επιτροπής. Δεύτερον, ανταγωνισμός, δίκαιος ανταγωνισμός. Η Επίτροπος Βιενκόσκα είναι η υπεύθυνη για, την, ε, για τον ανταγωνισμό, το δίκαιο ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αυτός ο δίκαιο ανταγωνισμός για τι εταιρείε οι οποίες συμμορφώνονται με τον κανονισμό ο οποίο ίσχυε το 2007. Και τώρα οι εταιρείε θα ακούνε πως οι ανταγωνιστέ του που δεν συμμορφώνονται θα λάβουν 5, 6, 7 χρόνια για να συμμορφωθούν επιπλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα εδώ ανταγωνισμού, δίκαιο ανταγωνισμού. Νομίζω ότι δεν είναι άδικος και ότι αλλάζουν οι κανόνες την ώρα του παιχνιδιού. Τρίτον. Μα είπατε πω τελικά συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θέλησε να αποφασιστεί το θέμα σύντομα και να μην χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Αν κατάλαβα καλά όμω, δεν συμβαίνουν και πολλά από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Αλλά εντάξει, κάποια δοκιμαστικά στάδια με δοκιμές για τις εκπομπές, αλλά με την περιορισμένη γνώση του θέματος που έχω, νομίζω ότι έφτανε ο χρόνος για να δώσει τη μάχη υπέρ των δικών της προτάσεως η Κομισιόν. Σχολιάστε το αυτό παρακαλώ. Τέλος. Κάτι το οποίο δεν κατάλαβα καθόλου. Τι θα συμβεί από τώρα και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 γιατί έχουμε τις παλιές ε, μεθόδους ε, δοκιμών και θα ξεκινήσετε εσείς με κάποιες πιλωτικές ε, δοκιμές για τις εκπομπές, δηλαδή δύο διαφορετικές δοκιμές με δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτά τα διαφορετικά αποτελέσματα θα δημοσιεύονται. Εμείς ως πολιτικοί και ακόμα πιο σημαντικό ως καταναλωτές, σε αυτά τα δύο χρόνια Πώς θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των πραγματικών εκπομπών και των εργασιακών δοκιμών. Δηλαδή πιστεύετε ότι για δύο χρόνια αυτή είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να κρατήσει και να διαρκέσει για δύο ολόκληρα χρόνια. Είναι πολύ τεχνικό και αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκίρλινγκ έχει το λόγο. Ξέρουμε όλοι πως το 2011 η DG Growth ξεκίνησε τις προσπάθειες να δημιουργήσει αυτές τις δοκιμές. Είχαν άλλο όνομα τότε, αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν η προσπάθεια που έκαναν, γιατί ήξεραν πολύ καλά ποιες είναι οι δυσκολίες και οι περιορισμοί του συστήματος που έχουμε στήσει και πως τα οχήματα πραγματικά δεν συμμορφώνονται με τον ε, περιορισμό στις εκπομπές. Το 2014 η Τεχνική Επιτροπή έφτασε σε ένα σχέδιο συμφωνίας, τουλάχιστον στο πρώτο τμήμα, το, το δεύτερο τμήμα της συμφωνίας το είδαμε μόλις την περασμένη εβδομάδα και αντιμετωπίζουμε σήμερα μία, ένα συμβιβασμό που δεν είναι ιδανικός. μα ζητάτε μία μεταβατική περίοδο για τον κύκλο ζωής των οχημάτων. Ε, εντάξει, λογικό, αλλά δεν καταλαβαίνω και θέλω εδώ να μου το εξηγήσετε πώς οι τιμές κατά τη διάρκεια της μεταβατικής, τιμής, μεταβατικής περίοδου με αποφασίστηκαν. Από πού προκύπτουν ή απλώς αποτελούν ε, τμήμα μιας ε, δημοπρασίας ή μιας ανταλλαγής που έγινε στην Επιστημονική Επιτροπή. Και για τα νέα οχήματα έχουμε κάποια σχέδια για να επιταχύνουμε την παραγωγή τους. Έχουμε ε, μελέτη για το κόστος των οχημάτων αυτών είναι λογικό και το κόστος να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια λήψης απόφασης. Αλλά γιατί δεν γίνεται με διάφορο τρόπο. Φαίνεται μάλλον ασαφές το τοπίο και εδώ. Όταν μιλάμε για μια διακοπή της διαδικασίας ή μια επιβράνευση της διαδικασίας, ε, εμένα δεν θα μου βρείτε σύμφωνη. Εγώ θέλω ίσα ίσα να επιταχύνουμε. Χρειαζόμαστε για τις αστικές περιοχές κυρίως πιο καθαρό αέρα το συντομότερο δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη του Κοινοβούλιο, οι κατασκευαστές συμφωνούν. Και όποιος παριστάνει πως πριν από τις αποκαλύψεις δεν είχαμε γνώση του προβλήματος με τις εκπομπές, πρέπει να ζει σε άλλο πλανήτη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι επειδή δείχνουμε τώρα μία θέρμη για να φτιάξουμε την κατάσταση, δεν μιλάμε με αυτούς οι οποίοι πραγματικά πλήττονται και μιλώ για ολόκληρη την οικονομία που ζει από την κατασκευή αυτοκινήτων, μιλώ για τους αυτο κινητοβιομηχάνους, αλλά μιλάω για τους εργαζόμενους σε αυτή τη βιομηχανία, γιατί ξέρετε πως η αυτοκινητοβιομηχανία είναι κινητήριος μοχλός για την απασχόληση στην Ευρώπη, όπως επίσης και για την πράσινη απασχόληση. Δεν θέλω λοιπόν να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου εμείς θα αρχίσουμε να κυνηγάμε αυτό τον εύκολο στόχο και τελικά να μην το αντιμετωπίσουμε παρά μόνο να δημιουργήσουμε όλο και περισσότερο προγράμματα ε, να πληγεί η βιομηχανία και να μην φτιάξουμε αυτή τη νέα τεχνολογία η οποία είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε το πρασίνισμα ε, της Ευρώπης. Thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ. Μια πρώτη ε, αντίδραση στη συνάδελφο. Εύκολος στόχος. Ε, δεν νομίζω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί έναν εύκολο στόχο. Ήταν πολύ αποτελεσματική στο να καθυστερεί τη δράση μας και στο να εξασφαλίζει πως οι στόχοι του οποίου θα πρέπει να πετύχουν παρατείνονται, καθυστερούν και πάλι και μάλλον ε, αποδυναμώνονται κιόλα. Γιατί αν είσαι εύκολο στόχο, αναρωτιέμαι γιατί στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, εκεί τα όρια είναι δύο φορές πιο αυστηρά και ίσως και πολύ πιο αυστηρά στην Καλιφόρνια, ενώ η Ευρώπη το 2006 μιλούσε για το 80, ενώ στην Καλιφόρνια έχουν ε, όριο το 35. Άρα λοιπόν μην τους λέτε και εύκολο στόχο. Εδώ συζητάμε αυτές τις πραγματικές δοκιμές. Να σας πω πως καταρχήν χαίρομαι που επιτέλους έχουμε μια νέα δοκιμή, η οποία ανακοινώθηκε όταν είχαμε συμφωνήσει το Euro 6, δηλαδή 8 χρόνια μετά τη συμφωνία, επιτέλους έχουμε και τη δοκιμαστική μέθοδο που χρειάζεται. Αλλά δεν είμαι καθόλου πεπισμένος και τελώ σε απόλυτη σύγχυση γιατί θα τους δώσουμε επιπλέον χρόνο έτσι ώστε να πλησιάσουν ένα όριο το οποίο εμείς συμφώνησαμε το 2007. Και Έχω και κάποια σημεία που είναι πολύ προβληματικά και νομίζω ότι σε νομικό επίπεδο είναι προβληματικά και αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από όλη τη στην οποία ανήκει ο καθένα μα. Πρώτα απ' όλα, μεταβατική περίοδος. Τα επιχειρήματα λένε πως η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να υιοθετήσει αυτέ τις νέε δοκιμέ. Προσπαθούμε απλώ να καθυστερήσουμε μία προθεσμία η οποία έχει θεσπιστεί για να πετύχουμε αυτό το όριο που είναι το 80. Δηλαδή, μεταβατική περίοδος, όταν ξέρανε ότι θα γίνουν αυτές οι δοκιμές, γιατί έχουν συζητήσει γύρω από ένα τραπέζι αυτές τις δοκιμές, για ποιο λόγο χορηγείται. Σε νομική βάση και μέσω της επιτροπολογίας πώς το δικαιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί να καθυστερούμε την εφαρμογή ενός ορίου που αποφασίσαμε το 2007 και θα έπρεπε ήδη να έχουν πετύχει το 2014. Δηλαδή επιπλέον χρόνο τι είναι αυτές οι νέες δοκιμές. Είναι μια έκπληξη που έσκασε μπροστά μας. Όλοι ήξεραν και διαπραγματευόντουσαν αυτές οι νέες δοκιμαστικές μεθόδους. Πού είναι η επιτροπολογία που τους οδηγεί στο να τους χορηγηθεί αυτή η μεταβατική περίοδος. Και μετά λέμε πως υπάρχει αυτό παράγον συμμόρφωσης που ουσιαστικά αποδυναμώνει το στόχο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μια εξαιρετικά δυσνόητη εξήγηση από πού προέρχεται, έχουμε δηλαδή το στατιστικό σφάλμα κτλ. Αλλά ξέρετε, εμείς το συζητήσαμε με την ε, Επίτροπο κυρία Μπιανκόφσκα και αυτή μας εξήγησε πού βασίζεται το στατιστικό λάθος στην πρόταση της Κομισιόν όπου κατέληξαν σε ένα παράγοντα 1,18. Τι σημαίνει 1,18 μακροπρόθεσμα. Πάντω αυτό που μα έχετε βάλει στο τραπέζι τώρα είναι το 1,5. Δηλαδή σε διαδικασία επιτροπολογία έχουμε θεσπίσει νέο στόχο. Με το 120 πια. Δεν συζητάμε πια το 80 ω όριο, αλλά το 120. Και αυτό είναι νέο στόχο Έχει νομοθετηθεί από το 2007 και αποδυναμώνεται και το αλλάζεται μέσω επιτροπολογία. Αυτό είναι απαράδεκτο απαράδεκτο για οποιαδήποτε πολιτική ομάδα. Δηλαδή εδώ δημιουργούμε ένα προηγούμενο όπου η επιτροπολογία χρησιμοποιείται και είναι μια τεχνική φύση διαδικασία, χρησιμοποιείται για να καθυστερήσουμε και να αποδυναμώσουμε στόχο τον οποίο έχουμε συμφωνήσει από το 7. Και αυτό είναι κάτι ε, το οποίο αναγνωρίζει η ίδια η Κομισιόν. Με το στατιστικό λάθος λοιπόν θα έπρεπε να φτάσουμε το 1,18 αυτό το 1,5 είναι πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση, πολιτικές ανταλλαγές οι οποίες δεν θα πρέπει να συμβαίνουν στη διαδικασία επιτροπολογίας και αυτό το κοινοβούλιο θα πρέπει να το περιγράψει ε, ανοιχτά και να τραβήξει μια γραμμή και να πει αν θέλετε κάτι τέτοιο θα το κάνουμε νομοθετικά ως συνομοθέτης και όχι εσείς μέσω επιτροπολογίας. Διαφορετικά ε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ευχαριστούμε κυρία Πύρικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη πολλές ερωτήσεις έχουν ε, αγιορθεί. Εγώ θυμάμαι την πρώτη συνομιλία που είχαμε εδώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλήσαμε για τον κανονισμό των ε, πραγματικών δοκιμών, των δοκιμών σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης. που πολύ συχνά συνδέονται με το θέμα της Ευρωπαϊκής Αποπτικής Αρχής στο Στρασβούργο. Το Κοινοβούλιο πέτυχε να εγκριθεί ε, η σχετική απόφαση και παρόλα αυτά το θέμα δεν έχει προχωρήσει. Εδώ μιλούμε για ε, άδειε, αδειοδότηση και εξουσιοδότηση σε κάποιου τομεί. Υπάρχουν περισσότερα περιθώρια από τις άλλους. Ε, επίσης αναμένουμε την διάσκεψη των μερών στο Παρίσι, την ε, διεθνή διάσκεψη. Και βάσει αυτής της προοπτικής είχαμε αποφασίσει ότι θα εξετάσουμε τα δύο θέματα σε ισότιμα. Ότι θα υπολογίσουμε τα μιλιγράμμ στον ε, τομέα της χαλιβουργίας, ε, το ίδιο και στον γεωργικό, την ε, ευζοία των ζώων, αλλά δεν είμαστε αρκετά ε, λεπτομερείς εδώ στις λεπτομέρειες. Ήμουν διακοπές την περασμένη εβδομάδα και έμεινα στην εκλογική μου περιφέρεια, σπίτι μου. Μίλησα με πολλούς εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας και μου, λένε, ε, και μου λέγαν ότι φαίνεται πολλά πράγματα να συμβαίνουν στο κοινοβούλιο, αλλά εγώ όσο βρίσκομαι εδώ θα, συζητάω, να, ε, θα συνεχίσω να ζητώ ίσους κανόνες για όλους. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε εδώ σήμερα και μα είπε ότι χρειάστηκε ένα συμβιβασμό. Όμω, κατά την άποψή μου, αυτό δεν είναι καν συμβιβασμό. Πριν από 8 χρόνια αποφάσισε 8 μιλιγκράμμα, 80 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, τώρα μα λέτε ότι συμβαστήκατε και αποφασίσατε 1,68 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο. Τι συμβασμό είναι αυτό, αυτό δεν είναι καν συμβασμό. Εάν πριν από 8 χρόνια αποφασίσαμε 80 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρα, πώ τολμάτε να μα λέτε ότι ήρθατε εδώ ε, και να μας λέτε ότι εγκρίνεται 168 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο επειδή συμβαστήκατε. Και αν δούμε τι έγινε και το 2007, το άρθρο 5.1 του κανονισμού Euro 6 είναι πολύ σαφές. Λέει 80 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο για τα οξύδια του αζότου πρέπει να επιτευχθεί ως στόχος της ε, ε, πραγματικέ συνθήκε οδήγηση. Δεν αναφέρεται καμία ευελιξία και κανένα περιθώριο σφάλματο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε και ανέφερε επακριβώ τον όρο ευελιξία. Μα είπε ότι χρειάζεται ευελιξία 1,8% για το 2019 και ευελιξία ε, του 15% ε, μέχρι το 2020. Αυτό που μας λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι είναι, ποια είναι η νομική βάση επί της οποίας η, Επιτροπή, η Τεχνική Επιτροπή αποφάσισε να αλλάξει τα όρια. Η αρχική νομοθετική πρόταση δεν αναφέρει καμία δυνατότητα ευελιξίας. Και δεύτερη ερώτηση. Εάν δούμε την περίοδο μετά το 2020, ο αριθμός 1,5 αντίκειται τελείως στην ίδια την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ό,τι μόλις ακούσαμε. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, παράγοντα συμμόρφωσης ε, συμβατότητας ε, με καταμέτρηση στο βαθμό 1,2%. Πώς φτάσατε τώρα στο 1,5% κάτι που αντιφάσκει με τη δική σας την αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν σημαντικό να ξέρουμε οι μελέτες και τα αποδεκτικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οδήγησαν στο 1,5% για μετά το 2020. Και η τελική μου ερώτηση θα ήθελα ε, ε, λεπτομερή παρουσίαση για τα αίτια που σας οδήγησαν να ε, να ε, επιτρέψει στην αυτοκινητοβιομηχανία να μισεύεται τα όρια που είχαν συμφωνηθεί πριν από νοκταετία. Έχουμε πει επανειλημμένω ότι οι τεχνολογικέ λύσει για να πετύχουμε τα όρια του Euro 6 ε, είναι διαθέσιμε. Δεν ισχύουν, δεν είναι και τόσο δαπανηρή λύση συνήθω. Εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι λέτε γι' αυτό. Υπάρχουν οχήματα που έχουν ήδη πετύχει το όριο του 80 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο. Ίσως έχετε εδώ κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Αν όμως δεν έχουμε τέτοιες χειροπιαστές απαντήσεις, καταλήγουμε στο, ε, σε ένα λογικό συμπέρασμα που δεν θα ήταν και τόσο ε, ευχάριστο. Ευχαριστούμε κυρία Μπέρντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι σχεδόν εισηγήτρια για την ε, πρόταση την νομοθετική πρόταση που εγκρίναμε στην ε, ε, Ολομέλεια τον περασμένο μήνα. Ο Επιτρόπος Βέλλα της συζήτηση στην Ολομέλεια είπε ότι όλοι οι τομεί θα πρέπει να έχουν το ίδιο φορτίο, ε, την ίδια το ίδιο μερίδιο ευθύνη στην πορεία προς καθαρή ατμόσφαιρα. και ότι θα πρέπει όλα τα κράτη να πετύχουν τα ίδια ε, εθνικά όρια. Όμως οι πόλεις και οι χώρες έχουν αποτύχει εξαιτία των εκπομπών ε, οξυδίου του αζότου κατά κύριο λόγο και κυρίως λόγω των οχημάτων diesel. Τον Σεπτέμβριο ε, βρέθηκε από μελέτη ότι μόνο ένα στα δέκα από τα ευρωπαϊκά οχήματα πέτυχαν τον, το όριο των 80 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο στις πραγματικές συνθήκες οδήγηση οδήγησης. Τώρα ο κανονισμός γύρω 6 όπως αναθεωρείται θα επιτρέπει διπλασιασμό των ορίων που ισχύουν σήμερα και 50% παραπάνω από το 2020 και πραγματικά με τρόμο διαπιστώνω ότι η Βρετανική κυβέρνηση η ίδια, η κυβέρνηση της χώρας μου δέχτηκε την αποδυνάμωση των ε, δοκιμών σε συνθήκε πραγματική οδήγηση. Το βρίσκω σκανδαλώδε διότι πραγματικά προκαλούνται θάνατοι και ε, χάνονται ζωέ και υπάρχουν απώλειες για όλες τις κοινότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός λοιπόν ο παράγοντας συμβατότητας 1,5% πώς ε, θα ε, εφαρμοστεί, πώς θα πετύχουν τα όρια οξυδίου του αζότου και των εκπομπών τους ε, τα κάτι μέλη, ενώ υπάρχει και ο παράγοντας συμβατότητας 1. Επίσης είναι σκόπιμη η πρόταση αυτή, είναι αρκετά αυστηρή με τα φορτηγά και τα λεωφορεία συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την στόχο να μειώσει κατά 52% του θανάτους από την κακή ατμόσφαιρα έως το 2020. Και έπειτα στο ανακοινωθέν σας στον τύπο χρησιμοποίησατε τον όρο κατά μεγάλο βαθμό να αποφευθεί παραποίηση μέσω συσκευών. Αυτό είναι το επίπεδο φιλοδοξιών που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θέλετε απλώς να περιορίσετε την παραποίηση ή απλώς να την πάψετε, να την καταργήσετε θα πρέπει ε, ο ατμοσφαιρικός αέρας που αναπνέουν οι πολίτες της πόλης να είναι όσο το δυνατόν ε, ποιοτικότερος και καλύτερος. Δηλαδή ότι ορίζεται το, το Euro 6. Το Euro 6. Ευχαριστούμε ο Αντιπρόεδρος Γιάβορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που δεν άκουσα να συζητείτε σε όλη αυτή τη συζήτηση ήταν να γίνεται κουβέντα ξεκάθαρη Ακούσαμε νούμερα, αριθμούς, ποσοστά, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα παράγοντα συμμόρφωσης, 2,1, που προτείνει το Συμβούλιο. Και συμφωνώ με τον Ματία Χρότα ότι πρόκειται για μια γελία κατάσταση, για πρόκειται για ανέκδοτο, δεν είναι παράγον συμμόρφωσης. Ουσιαστικά σημαίνει οπισθοδρόμηση σε σχέση με τον παράγοντα με τις προδιαγραφές ε, Euro, 5, Euro 6. Πάμε πίσω στις Euro 5. Νομίζω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει μια πρόταση η οποία να μιλάει ξεκάθαρα για τις προθέσεις της Επιτροπής και να μην ε, μας ε, ξεγελάνε με παράγοντες συμμόρφωσες. Από την άλλη νομίζω ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκηνικό θεάτρου. Ενοχλούμαστε βέβαια και προσβαλόμαστε για το παράγοντα 2-1 και τα λοιπά Παράγοντα μόρφωσης. Σαν να είμαστε σε μια ταυρομαχία και να μας κουράνε το κόκκινο πανήμα. Αυτό ακριβώς για αυτό το λόγο γίνεται, για να ε, συγκεντρώσουμε τις επιθέσεις μας στον παράγοντα συμμόρφωσης 2-1, γιατί αρχικά είχε στήσει 1,6 η Επιτροπή. Παράγοντα μόρφωση, που επίσης είναι γελίο. Και για να εξηγήσω καλύτερα, από άποψη τεχνική, ο παράγοντας μόρφωση δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση οικονομικών ή προβλημάτων παραγωγή βιομηχανική, αλλά με την αβεβαιότητα σε σχέση με κάποιε μετρήσει. Παράγοντας συμμόρφωση 1,2 που αποδεδειγμένα προκύπτει από τις μελέτες. Οτιδήποτε λοιπόν ξεπερνάει το 1,2 και πάει στο 2,1 κτλ, είναι πολιτική επιλογή και όχι τεχνική. Πολύ φοβούμαι λοιπόν ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι το Κοινοβούλιο θα αντιδράσει στον παράγοντα συμμορφώσεις 2-1, μεγάλη έμφαση, για να καταλήξουμε σε μια ωραία συμβαστική λύση της τάξης του 1,6, που τελικά είναι αυτό που θέλουν να επιτύχουν οι άλλοι. Και άρα ανατρέπει οτιδήποτε κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι πέραν του να διατυπώνουμε τις επικρίσεις μας για την πρόταση αυτή του 2,1 που συμφωνούμε πιστεύω όλοι οι περισσότεροι, δεν πρέπει και να δεσμονούμε πως συμβασμός στο 1,6 οποιοδήποτε άλλο συμβασμός τέτοιου τύπου θα είναι πάλι πολιτική απόφαση και δεν έχει καμία σχέση με τεχνικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Προς τον ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής θα παραθέσω τις ε, παρατηρήσεις της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου που λέει ότι σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσεως πρέπει να τηρούνται οι όροι του Euro 6 πρώτον. Δεύτερον, δεν αφισβητούνται οι κανόνες συμμόρφωσης από το Κοινοβούλιο, αλλά ο τρόπος εφαρμογής. Και η νομική υπηρεσία ξεκάθαρα τοποθετείται με την αξιολόγηση και την ανάλυση της αποφάσεως της προηγούμενης εβδομάδας και μας λέει ότι το δεύτερο σχέδιο κανονισμού που εξέτασαν οι πυρογνώμονες των κρατών μελών θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ξεπερνά την εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους όρους εξουσιοδότησης. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή πώς σκοπεύει να προχωρήσει από εδώ και μπρος. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Επιτροπή, εκτό βέβαια και αν ε, παρισφρήσει απόφαση σε επίπεδο τεχνικό και από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ε, πώς ε, θα προχωρήσει λοιπόν από εδώ και μπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παραγνωρίσει τις ε, αποφάσει του Κοινοβουλίου. Και δεύτερον, για να επανέλθω με μια ερώτηση που είπε η κυρία Σράιερ νωρίτερα, είναι ο τύπος της εγκρίσεως με μια απόφαση του Κοινοβουλίου πριν από δύο εβδομάδες που δηλώνει ξεκάθαρα και η κυρία Πιανικόφσκα φαντάζομαι θα είχε το χρόνο να τη διαβάσει μεταξύ για την προηγούμενη εβδομάδα την επιβέωση Ρωτώ λοιπόν τον εκπρόσωπο της Επιτροπής εάν όντως αυτές είναι οι προθέσεις της Επιτροπής να καταθέσει δηλαδή πρόταση για μια εύρωστη ευρωπαϊκή εποπτεία των εγκρίσεων εθνικού τύπου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάνς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την αίσθηση ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζανε πως το θέμα αυτό θα εξαφανιστεί, ότι δηλαδή δεν θα το συζητάμε πια και ότι αν κάπως ε, χαϊδολογήσουμε τους στόχους θα αλλάξουν. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί το θέμα μέχρι να καθαρίσει ο αέρας που εισπνέουμε. Είναι ένα πολύ ε, συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι αφηρημένο, είναι ε, ουσίες που ρηπαίνουν το περιβάλλον που κυκλοφορούν στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συναπόφασης και πριν από 8 χρόνια συναπόφαση θέσπισε πολύ αυστηρούς ε, όρους για ε, πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ποια είναι η νομική βάση για να αλλάξει αυτός ο στόχος μέσω επιτροπολογίας. Και αν ο στόχος δεν είναι να αλλάξει, μάλλον αν η προσπάθεια δεν είναι να αλλάξει ο στόχος, αλλά απλώς να αλλάξουμε το παράγοντα συμμόρφωσης προς το 1,5, πώς θα λειτουργήσει. Γιατί το 1,5 επί το 80 νομίζω θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα υψηλότερο του 80. Αν κάνει κανείς τον πολλαπλωσιασμό φαντάζομαι. Ε, πείτε μου λοιπόν τι θα συμβεί. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. βλέπω εδώ μια αλλαγή επιχειρηματολογίας και έχουμε ξαναρωτήσει και στο παρελθόν, συζητάμε εδώ την αλλαγή των στατιστικών, πώ προσπαθούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Μάλλον φαίνεται ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την πραγματικότητα και όχι να αλλάξουμε τις στατιστικές. Στις στατιστικές, στο εργαστήριο δηλαδή, έχουμε κερδίσει ήδη τη μάχη από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχουμε πρόβλημα με την πραγματικότητα και πρέπει να την αλλάξουμε και αυτήν. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή. Πρώτον, Υπάρχει κάποια γενική εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση στην πραγματικότητα. Πληρούνται οι όροι του Euro 5 ή πώς θα πέσουμε και στο Euro 4 τελικά. Ποια είναι η πραγματικότητα. Ή να το πω διαφορετικά, ποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές μπορούμε τελικά να τηρήσουμε έτσι όπως έχει η κατάσταση και αν είναι να βελτιώσουμε την ε, πραγματικότητα, ε, α ορίσουμε και πιο ρεαλιστικούς στόχους, δηλαδή στόχους που μπορούν να τηρηθούν. Και άλλη μια ερώτηση προς εμάς. Κυρία Σάιρ Πύρικ το είπε και νωρίτερα. Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουμε τα πραγματικά δεδομένα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η οδηγία για τις ε, εκπομπές. και να ορίσουμε έτσι και πιο ρεαλιστικούς στόχους για τη γεωργία και να κοιτάξουμε τι άλλη βελτίωση χρειάζεται στις μεθόδους αλλά και στους στόχους. Πρέπει ίσως να το ξανακοιτάξουμε αυτό το θέμα της οδηγίας και να την ξαναδιαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ακούσατε πολλά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. για την πρώτη ερώτηση που είναι τα κείμενα. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι μεταφράσεις και η ημερομηνία που μας δόθηκε είναι 23η Νοεμβρίου. Οπότε θα έχουμε έτοιμες όλες τις μεταφράσεις και θα μπορούμε να σας στείλουμε όλα τα κείμενα αυτά. Δεύτερον, αν κατάλαβα, εάν η πρόταση μπορεί να τροποποιηθεί Ξέρετε πως η αρχική μας πρόταση ήταν ε, διαθέσιμη και βεβαίω ε, σχολιάζουν τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή και μπορούν να τροποποιήσουν αν είναι μια πλειοψηφία κρατών μελών που το επιθυμεί. Ο κύριος Φλόρεντς μίλησε για τις επιπτώσεις. Να σας πω πως ε, οι κατασκευαστές μας λένε πως τα αποτελέσματα της Τεχνικής Επιτροπής για τα αυτοκίνητα οχήματα λένε πως το 30 με 50% των ε, υφιστάμενων οχημάτων θα πρέπει να προσαρμοστούν για να ε, μιλάω για τα ντίζελ, εντάξει, πετρελαιοκίνητα θα πρέπει να προσαρμοστούν για να συμμορφωθούν με τις ε, επιταγές της νομοθεσίας. Για το διοξίδιο του άνθρακα θα αφήσω το συνάδελφο να απαντήσει. Μια δεύτερη ερώτηση από σας άκουσα και για την νομοθεσία. Νομίζω πως το γεγονό πως εισάγουμε αυτές τις πραγματικές δοκιμές κάνει πιο συγκεκριμένη την νομοθεσία. Όπως σας υπενθύμησα, οι πραγματικές εκπομπές σε σχέση με τις πραγματικές δοκιμές είναι κατά μέσο όρο τέσσερις φορές υψηλότερες. Το γεγονός λοιπόν πως εισάγουμε είναι απόδειξη πως εφαρμόζουμε πιο σωστά την νομοθεσία. Η Επίτροπος Βιενκόφσκα είπε πως αυτή τη στιγμή αναθεωρούμε την διαδικασία έγκρισης τύπου και το πιο ουσιαστικό στοιχείο είναι αυτό, γιατί θα επιτρέψει την νομοθεσία να εφαρμόζεται πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά, να γίνεται περισσότερο σεβαστή. Είχαμε βέβαια κάποιους στόχους αρχικά, και είχαμε και διάφορες λίτρες ε, διασφάλισης, ρήτρες απόσυρσης, επιτήρηση από την, και παρακολούθηση από την Κομισιόν. Αυτό το βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά τώρα βέβαια και υπό το φως των ε, γεγονότων. Με το γεγονός αυτό λοιπόν οδηγηθήκαμε στο να ε, εφαρμόσουμε πιο αυστηρά και πιο γρήγορα κάτι το οποίο είχαμε ήδη κατά νου. κύριος Καπράνη και τα σχόλιά τους, δεν θα μιλήσω για τα ανακοινοθέντα τύπου και για το κατά πόσο ήταν σωστός ο τόνος μας. Πάντως στην πράξη οι εκπομπές πρώτα θα μειωθούν κατά το ίμιση τουλάχιστον και στο τέλος της διαδικασίας νομίζω ε, στην πράξη θα είναι τέσσερις φορές λιγότερες. Θέλω να θυμόσαστε πως εάν δεν εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τα όρια των πραγματικών δοκιμών, θα οδηγήσουν στο να μείνουμε με την τρέχουσα κατάσταση, η οποία είναι 400 ανά χιλιόμετρο. Μιλιγκράμμα ανά χιλιόμετρο. Τώρα, ανταγωνισμός. Δίκαιος ανταγωνισμός. Το γεγονός πως η αυτοκίνητο βιομηχανία σέβεται την τρέχουσα νομοθεσία δεν σημαίνει πως στην πράκτη ε, σε πραγματική χρήση εφαρμόζει τους στόχους που είχαμε. Και αυτό ήταν το πρόβλημα των εργαστηριακών δοκιμών. Όπως σας είπα είναι τέσσερις φορές παραπάνω από ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, το ότι ένα όχημα συμμορφώνεται με την ε, νομοθεσία δεν σημαίνει πως σε οδική, σε, ε, ε σε εκπομπές πραγματικές εν ώρα οδήγησης σέβεται το στόχο που είχαμε θεσπίσει ως όριο. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τι θα συμβεί μέχρι το 2017 από σήμερα. Οι νέες δοκιμές θα είναι συμπληρωματικές στις παλιές Γίνονται ήδη τα πιλωτικά, αλλά για την 1η Ιανουαρίου του 2016 θα χρησιμοποιηθούν οι δοκιμές αυτές και για στόχους παρακολούθησης, έτσι ώστε αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων να καλυφθεί. Αυτό θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση της κατάστασης και ίσως τον παράγοντα συμμόρφωσης να τον ανανεώνουμε σε αιτήσια βάση. Και αυτό θα μας δώσει μια βάση για να γνωρίζουμε πιο συγκεκριμένα ποιο είναι ο παράγοντας συμμόρφωσης που χρειάζεται. Πώς καταλήξαμε σε αυτές τις τιμές. Βασιζόμαστε καταρχήν στις ίδιες τις δοκιμές, στη μεθοδολογία δηλαδή, και δεύτερον η αβεβαιότητα με τα αποτελέσματα τα οποία θα δώσουν οι δοκιμές ε, σε πραγματικές συνθήκες. Γιατί εξαρτάται βέβαια από την κλίση του δρόμου στον οποίο θα γίνουν οι δοκιμές, από την επιτάχυνση για παράδειγμα. Οπότε έχουμε πει πως αυτός ο παράγοντας συμμόρφωσης θα πρέπει να ακολουθεί μια υψηλότερη τιμή και εδώ έχει το αποτέλεσμα του συμβιβασμού. Έχουμε και ρήτρα αναθεώρησης, γιατί όσο πιο πολύ έχει προχωρήσει η εφαρμογή αυτών των νέων δοκιμών, τόσο πιο πολλά θα γνωρίζουμε. Και μετά θα μπορούμε να προσαρμόσουμε και αυτόν τον ε, συντελεστή. για τις ε, πιο αυστηρές ε, διατάξεις ε, στη ΣΥΠΑ και για τα όρια εκεί δεν έχουν πετρελαιοκίνητα στην Αμερική. Και τα δικά τους επίπεδα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξα από τα δικά μας. Για τον όρο flexibility, περιθώριο λιγμών ουσιαστικά να σε εξηγήσω για το συντελεστή λοιπόν αυτό συμμόρφωσης, να σας πω ακριβώς ε, τι συμβαίνει. Δεν είναι ευέλιξη για να είμαστε ευέλιξοι, είναι ένα περιθώριο που δίνουμε, μια ανοχή, λόγω της αβεβαιότητας και της διαδικασίας και του τρόπου που θα εφαρμόζεται η δοκιμή και αυτό το περιθώριο σκεφτήκαμε πως θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού και έτσι καταλήξαμε σε αυτή την τιμή. Πώς συνδέεται βέβαια με το συντελεστή συμμόρφωσης ε, ποιότητας ε, ατμοσφαιρικού αέρα δεν συνδέονται τα δύο αυτά γιατί ο ατμοσφαιρικός αέρας ε, υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκπομπές πάντως η επίπτωση των εκπομπών οξυδίων αζότου επηρεάζει βέβαια και τα δικά μας όρια παρόλο που με τις πραγματικές δοκιμές θα καταλήξουμε σε ένα συντελιστή που είναι πολύ χαμηλότερος από τον τρέχοντα. Ουσιαστικά 24 μιλιγραμμ ανά χιλιόμετρο, κάτι το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς όντως θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν κάτι να μου υποδείξουν. Ξέχασα κάποιον. Για το πώς θα συνεχίσουμε εάν το Κοινοβούλιο θεωρήσει πως έχουμε υπερβεί τα εσκεμένα. Νομίζω αυτό είναι δικό σας θέμα, εσείς θα αποφασίσετε. Και βεβαίως, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα σκεφτούμε και εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω αυτά είχα να πω. Φιλίπ, ίσως θες και εσύ να προσθέσεις κάτι. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα ζήτημα για το διοξείδιο του άνθρακα, μια ερώτηση. Μπορεί να κάνω και λάθος. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μάλλον θυμάστε καλύτερα από μένα. Θα ήταν μερικέ οι ερωτήσει για το δεξιό του άνθρακα. Ο κύριο Φλόρεντ, σε παράδειγμα, τη μίλησε για το κόστο συμμόρφωση με τι εκπομπέ οξυδίων του αζότου και αν ήταν συγκρίσιμο με αυτό των ε, οριακών τιμών για το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά δεν είμαι έτοιμο να δώσω απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Πολύ ευχαριστώ να το ξανακοιτάξω και να σα αποστείλω τι απαντήσει μου. Έχουμε βεβαίω καμπύλε κόστου ε, για το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά θα πρέπει να στου αδέρφου να κοιτάξουν ε, τη σύγκριση με το κόστο συμμόρφωση στα οξύδια του αζότου. Για το άλλο ερώτημα, το οποίο νομίζω αλλά την κατάσταση Ηνωμένε ΗΠΑ και νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκε ότι υπάρχουν προδιαγραφέ για το διοξείδιο του άνθρακα στις ΗΠΑ είναι δύσκολο να γίνει η σύγκριση βέβαια μεταξύ των στόλων ε, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της διαφοράς ε, στα μεγέθη, στους τύπους ε, των οχημάτων, τα είδη καυσίμων κτλ. Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές πάντως είναι ελαφρώς αυστηρότερες από τις αμερικανικές. Και ως προς το αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ οξυδίων του αζότου και διοξυδίου του άνθρακα, ιστορικά η απάντηση που δινόταν ήταν καταφατική, αλλά σιγά σιγά ε, δίνονται διαφοροποιήσεις σχέση με την βελτίωση της ποιότητας απόδοσης των κινητήρων πετρελαίου που μειώνουν αυτή τη διαφορά τα τελευταία χρόνια. Και πάλι έχουμε πληροφορίες στη θέση μας. Εάν ε, το επιθυμούν οι βουλευτές μπορώ να σας δώσω λεπτομερέστερε πληροφορίε. Καλώ. Ο κύριο Γκέρπραντι, μήπω θέλει κάτι να πει. Ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ρωτάω το εξή λοιπόν. Εάν κάθε εβδομάδα κλέβω από πέντε μήλα και με πιάσουν με πιάσει αστυνομία και προσπαθήσω να διαπραγματευτώ λέγοντα ότι α, από εδώ και προ εγώ θα κλέβω μόνο τρία μήλα. Για σας θεωρείτε ότι θα είναι μια τεράστια βελτίωση της καταστάσεως. That αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, η κατάσταση μεταξύ της κατάστασης όπως την έχουμε τώρα και εκείνης του θα του το του 2018 θα είναι ότι θα έχουμε δύο δοκιμές με αποτελέσματα στη διάθεσή μα, Όντως δύσκολη η διαχείριση της κατάστασης αλλά εσεί πάλι μιλάτε για 400 μιλιγκράμμ σε εκπομπές τώρα. Και άρα αυτό θα επιτρέπουμε για τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα έχουμε παράγοντα συμμόρφωσης πέντε για τα επόμενα τρία χρόνια. Καλά τα λέω. Ο Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί μου ζητούν το λόγο για συμπληρωματικές ερωτήσεις. Είναι προφανές ότι όλοι θέλουν να διατυπώσουν συμπληρωματικές ερωτήσεις. Να συνεχίσουμε αν θέλετε, αλλά τότε θα προτιμούσα να, κάνουμε, να ακουστεί μόνο μία ερώτηση και η συζήτηση να γίνει πιο ευρεία μια άλλη στιγμή. Ε, να προβλέψουμε καινούριο χρόνο, γιατί δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις που δόθηκαν. Πάντως βλέπω ότι όλοι έχουν διαμορφώσει άποψη για το θέμα. Και είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε και σε άλλα σε άλλε για συνάντηση με την Επιτροπή το θέμα αυτό. Δεν κλείνει σήμερα δηλαδή η συζήτηση. Και γι' αυτού του λόγου καλώ Του συναδέλφου να μην διατυπώσουν συμπληρωματικέ ερωτήσει γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και στο επόμενα θέμα τη ημερικής διάταξη. Αν θέλει να απαντήσει η Επιτροπή. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ να, θα προσπαθήσω να απαντήσω χωρίς να προξενήσω και άλλες ερωτήσεις. Για τα μήλα δεν θα σχολιάσω. Για το παράγοντα συμμόρφωση όμω θα ήθελα να σχολιάσω, γιατί δεν είναι, πραγματικ... δεν είναι σωστός ο τρόπος να παρουσιάζουμε την κατάσταση λέγοντας ότι έχουμε παράγοντα συμμόρφωσης 5, γιατί υπάρχει νομοθεσία και εφαρμόζονται οι δοκιμές. Ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα, για να έχει τη δυνατότητα να δια... διαθέσει ε, στην αγορά το όχημα που κατασκευάζει, πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις των προδιαγραφών και τις προδιαγραφές των δοκιμών και χωρίς βέβαια να έχουμε παραγόντα 5 όπως είπα, είμαστε πιο κοντά χάρη στις δοκιμές αυτές στην πραγματικότητα. Λόγω των αβεβαιοτήτων ε, ορίζονται και παράγοντες συμμόρφωσης. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι θα έχουμε παράγοντα συμμόρφωσης 5. Θέλουμε να κερδίσουμε μια εμπειρία με τις δοκιμές και βέβαια είναι απαραίτητη και η περίοδος μετάβασης για να μπορέσουν οι κατασκευαστές να προσαρμόσουν τα συστήματα παραγωγής κτλ. Θα ήταν άδικο νομίζω για την Επιτροπή να λέγεται πως ζητάει παραγωγές μόρφωσης 5. Καλώς λέει Πρόεδρος, κλείσουμε εδώ τη συζήτηση. Για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Στην ημερήσια διάταξη προφορική ερώτηση για την κατεργασία ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή ένωσε από των Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Ήταν ο κύριος Καλχάιντς Φλόρενς, εκείνος ο οποίος διατύπωσε την ερώτηση μαζί με τον κύριο Αικχάουτ και παρακαλώ και τους δύο ε, συντάκτες να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Φλόρενς. Ε, Χάιντς, με συγχωρείς ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε κλείσει τη συζήτηση για τις εκπομπές προς το παρόν. Παρακαλώ όμως, ε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το επόμενο θέμα, να μην ε, παρενοχλείτε. Χάινς Φλόρενς. Ναι. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη λεγόμενη κυκλική οικονομία, για τα τρία ε, ε για το κανονισμό. Δηλαδή, την ανάκτηση πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αξιοποιηθεί ήδη. Δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ε, κανονισμό για τα απόβλητα από ήδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ε, ο υποφαινόμενο και ο κύριος Εκχάτου τυπώσαμε αυτή την προφορική ερώτηση για να ρωτήσουμε την Επιτροπή τι, ε, τι έχει κάνει τελικά ε, για την ε, διασφάλιση της στήρησης των προδιαγραφών και των όρων του κανονισμού. Υπάρχουν βουνά παράνομα, παράνομου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπάζων ηλεκτρονικών, να το πω έτσι, μεγάλης αξίας, τα οποία διοχετεύονται χωρίς να, γίνεται, χωρίς να τηρούνται οι όροι της ε, απογύμνωσης από ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, δεν τηρούνται οι μελέτε, οι, οι όροι, όλα αυτά τα καταγράφει άλλωστε μια μελέτη και που επιβεβαιώνει τις υποψίες μας. Τη γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μελέτη και γι' αυτό την παρακαλώ να μας ενημερώσει για την κατάσταση. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε με τον Επίτροπο Βέλα για την κυκλική οικονομία, κυρίως εγώ. Και φτιάχνουμε έτσι ένα πολύ ωραίο μόρφωμα, όπου όμως πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν ε, και θα έπρεπε να δίνουν απαντήσεις στα ζητήματα του AAA, των ε, ε, αυτοκινήτων που δεν κυκλοφορούν πια, που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία και όλα αυτά, δεν τηρούνται. Και έτσι έρχεται μια, ένα νέο καταπληκτικό και όμορφο μόρφωμα για να δοθούν απαντήσεις σε πράγματα τα οποία όμως δεν υφίστανται. Γι' αυτό περιμένω από την Επιτροπή απαντήσεις. Ευχαριστούμε ο κύριο Σέκαουτ. Ο συνάδελφο Καρλ Χάιν το εξέφρασε άψογα στα γερμανικά. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω στα αγγλικά ή στα ολλανδικά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Γιούλιο Γκαρσία Μπέρκες που είναι επικεφαλής υπηρεσίας, διευθυντής υπηρεσίας και θα μας δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την προφορική σας ερώτηση και καλωσορίζουμε αυτή την ευκαιρία να την ανταλλάξουμε πληροφορίες για την αποκομιδή των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών δηλαδή. Πρόκειται για έναν αγοργά ε, αναπτυσσόμενο τομέα και από τη σκοπιά της κυκλικής οικονομίας μπορούμε να έχουμε μεγάλα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης. Είναι ένα θέμα με ευρύτατο πεδίο και οι πέντε υπερωτήσεις καλύπτουν ε, πολλά τα θέματα όπως το δεί κάνουμε με τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, την σχετική οδηγία WE και επίσης ε, το θέμα της υλοποίησής της και ούτω καθεξής. Θα απαντήσω ένα προς ένα και θα προσπαθήσω να είμαι ακριβής στις απαντήσεις μου, χωρίς όμως να αφήσω καμία ερώτηση αναπάντητη. Πρώτη ερώτηση. Τι συνέπειες προβλέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υλοποίηση της οδηγίας από την μελέτη SeaWit. Δεν είναι έκπληξη για μας τα πορίσματα της μελέτης SeaWit. Έχουμε έμεσες και άμεσες αποδείξεις που δείχνουν ότι σημαντικό ε, ποσό το, ε, των αποβλήτων αυτών είτε εξάγονται είτε τα διαχειρίζονται με το δικό τους τρόπο τα κρατημέλη. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι. Τα νομοθετικά εργαλεία υπάρχουν, ιδίω με την αναδιατύπωση της οδηγίας, αλλά πρέπει να ε, υλοποιηθούν ε, στην πράξη. Κατά πρώτον, η οδηγία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα προβλέπει συγκεκριμένε προϋποθέσεις για την ε, αποστολή των ε, εξοπλισμών που δεν λειτουργούν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Δίνει στους εθνικούς επιθεωρητές τις δυνατότητες να ε, μελετήσουν, να ε, ελέγξουν τις παρτίδες εάν θεωρήσουν ότι πρόκειται ενδεχομένως για παράνομη εξαγωγή αποβλήτων. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό εργαλείο, η αντιστροφή του παρός του βάρου απόδειξη μάλλον, και πρέπει ο κάτοχος ε, σε κάθε περίπτωση των αποκλήτων, κάτοχος του εξοπλισμού ε, αρχικά, να αποδείξει ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί και δεν πρόκειται για απόβλητο. Έπειτα, ο σχετικό κανονισμό τροποποιήθηκε πρόσφατα για να ενισχύσει τι διατάξει περί επιθεωρήσεων. Οι διατάξει που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου θα δώσουν περισσότερε εξουσίε στου ελεγκτές. Και επιπλέον, τα κράτη-μέλη θα καλούνται να προβλέψουν στην 1η Ιανουαρίου 2017 πρόγραμμα επιθεωρήσεων που θα πρέπει να βασίζεται σε αποτίμηση κινδύνου και να ορίζει ελάχιστο αριθμό ε, επιθεωρήσεων που θα πρέπει να διεξαχθούν. Ε, δεν χρειάζεται να διευκρινίσω ότι οτιδήποτε αφορά τους ελέγχους βρίσκεται στα χέρια των εθνικών αρχών. Τελωνιακές αρχές, επιθεωρητές αποβλήτων και αστυνομία. Ωστόσο, λαμβάνουμε και δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία συμμόρφωσης και ευθυγράμμισης ε, για την οδηγία GUI για να εντοπίσει στην πράξη τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την ε, ανακομιδή των ε, ανακυκλώσιμων και την καταπολέμηση της παρανόμης εξαγωγής. Κατά την υλοποίηση της, τη διεξαγωγή της πρωτοβουλίας αυτής θα συνεργαστούμε με το δίκτυο των Ευρωπαίων Περιβαλλοντικών Ελεγκτών που ήδη έχει ξεκινήσει πολλά προγράμματα για να αντιμετωπίσει τις λαθρές εξαγωγές αποβλήτων. Επίσης θα λάβουμε υπόψη τις σχετικές μας εμπειρίες για την ε, καθοδήγηση των υπευθύνων για την αναδιατύπωση της οδηγίας αυτής και τον καθορισμό των προγραμμάτων επιθεωρήσεων όπως προβλέπει η οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Συνεργαζόμαστε και με την Ιντερπόλ, από τους μεγαλύτερους εταίρους μας στο πρόγραμμα αυτό παγκοσμίω και συμμετέχουμε στην ομάδα εργασία για την καταπολέμηση των εγκλημάτων ρήπανση στο επίπεδο τη Ιντερπολ και σήμερα υπήρχε μια ημερίδα για τέτοιου είδου ε, λαθρέα διακίνηση, την οποία οργάνωσε η Ιντερπολ στο Βέλγιο. Επίση, είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε και τη διμερή συνεργασία και στηρίζουμε κάποια εγχειρήματα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων στι αναπτυσσόμενε χώρε και να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα ε, πρόγραμμα τελωνιακής συνεργασίας με την Κίνα, το οποίο επικεντρώνεται όλος ιδιαίτερα στις παρτίδες τέτοιου είδους αποβλήτων. Τέλος, θα δίνουμε τη συνεργασία μας με διεθνείς ε, φορείς και τις πρωτοβουλίες τους για την ανάπτυξη και υλοποίηση των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών, για την ε, μεταφορά των γουί, που ε, μελέτησαν οι συμβαλόμενοι στη Σύμβαση της Βασιλείας νωρίτερα φέτος. Τώρα για το δεύτερο σημείο, το πώς έχουν τα πράγματα ως προς την οδηγία και την υλοποίησή της από τα κάτι μέλη, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ποσοστά αποκομιδής, τους στόχους αποκατάστασης και τις επιθεωρήσεις, θα ήθελα να αναφέρω κατά πρώτον ότι οι τωρινοί στόχοι αποκομιδής, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας ΓΟΥΙ 40 κιλά ανακεφαλή εφαρμόζονται και η συνολική εικόνα δεν είναι κακή. Ε, η τελευταία χρονιά αναφορά, στο 2013, και παρόλο που κάποια, κάποια στοιχεία μας λείπουν ακόμη, βάσει των δεδομένων που έχουν ήδη υποπληθεί στη Eurostat, μόνον πέντε κράτη-μέλη δεν έχουν πετύχει τους στόχους συλλογής. Και κάποια από αυτά τα πέντε κράτη-μέλη είναι πολύ κοντά στο στόχο. Το επίπεδο συμμόρφωσης για τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης όπως ορίζονται στο παράδειγμα 5 της οδηγίας WE έχουν ε, λίγο πολύ επιτευχθεί αλλά όχι από τα κράτη-μέλη. Τρεις δεν τα κατάφεραν για τα αυτόματα μηχανήματα, και τα μηχανήματα επικοινωνίας. Ε, κάποιοι πρέπει να ε, προχωρήσουν ε, με, για τα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τις κατηγορίες αυτές προϊόντων. Για τις επιθεωρήσεις για το διάστημα 2012-2013 υπήρξαν τουλάχιστον 2.500 περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν παράνομες παρτίδες αποβλήτων βάσει των οποίων 50 ε, εκ των οποίων μάλλον 50% περίπου ήταν λαθρές αποστολές ε, τέτοιων αποβλήτων ηλεκτρολικών και ηλεκτρολογικών. Σίγουρα έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ε, λαθρέων αυτών αποστολών, αλλά αυτό δεν είναι αναγκαστικά μια αρνητική τάση. Δείχνει απλώς ότι οι επιθεωρήσεις γίνονται αποτελεσματικότερες και ότι ο και μεγαλύτερος αριθμός παράνομων αποστολών και παρτίδων εντοπίζονται. θα, θα απαντήσω από κοινού το ε, τρίτο και τέταρτο ερώτημα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ε, επίτευξη των στόχων περισσότερης ανακομιδής ε, όπω ορίστηκαν για το 2016, μα ε, ρωτούν στο τέταρτο ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει ε, μεγαλύτερα ποσοστά ανακομιδή στο στόχο για κάποιε κατηγορίε γουί. Θα τα απαντήσω από κοινού γιατί ξεκινήσαμε μια μελέτη όπου και τα δύο θέματα μελετήθηκαν εντελεχώς. Όσον αφορά την, το εφικτόν των ε, στόχων ανακομιδίου για το 2016 και ως το 2019, τα πορίσματα της μελέτης, η οποία ε, μόλις επιβιώθηκε, ακόμη δεν έχει καν δημοσιευθεί στον αστυτοπό μας, δείχνουν λοιπόν τα πορίσματα αυτά ότι κάποια κράτη-μέλη ίσως να μην είναι σε θέση να συμμορφωθούν πλήρως με τους στόχους, εάν δεν αντιμετωπίσουν κάποιες ανεπάρκειες στην υλοποίηση. Αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό των, ε, της ανακομιδής που δεν καταγράφεται ή την έλλειπη ε, ε, υλοποίηση κατά τις δυνατότητες παρακολούθησης. Η μελέτη εντοπίζει ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση σε 10 κατημέλη με ποσοστά ανακομιδής 2010 χαμηλότερα κατά 30% από την ανακομιδή Wii που είχε καταγραφεί την ίδια χρονιά. Αυτά τα κενά, αυτές οι ελλείψεις ε, στα κράτη-μέλη με τα χαμηλότερα ποσοστά ανακομιδής είναι ένα θέμα που θα το δούμε στην πρωτοβουλία για την πρόθεση της συμμόρφωσης. Κάτι που όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου θα ξεκινήσει του χρόνου. Η μελέτη επίσης αξιολογεί την δυνατότητα να ορίσουμε ξεχωριστούς ε, στόχους για ε, κάποιες ομάδες προϊόντων WE. Ε, ίσως αυτοί οι μονομένοι στόχοι να είναι πιο ωφέλιμοι από την από ή κοινωνικο-οικονομική Ε, είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τεθούν τέτοιοι στόχοι και να γίνουν σεβαστοί από τα κάτι μέλη. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι ίσως είναι αντιπαραγωγικό να ορίσουμε ξεχωριστούς στόχους ανακομιδής ενώ δεν έχουμε καν πετύχει τους ετήσιους στόχους ανακομιδής και δεν έχουν καν υλοποιηθεί για την ομάδα αυτή των προϊόντων WE η απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Υπάρχουν ξεχωριστές κατηγορίες προϊόντων λοιπόν και αν θέλουν τα κάτι μέλη μπορούν με δική του πρωτοβουλία να εφαρμόσουν ε, ξεχωριστούς στόχους αυτόνομους. Ίσως μια τέτοια μελέτη ήταν και ένα χρήσιμο εργαλείο για να στηρίξουμε την υλοποίηση ε, και την μελέτη επίτευξη των ετήσιων στόχων όπως τους ορίζει η οδηγία. Τελευταία ερώτηση. Πώς έχει η κατάσταση σήμερα σε σχέση με τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την ανακύκλωση. Συζητήσαμε με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης για να καταλήξουμε, τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης για να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές αυτά θα πρέπει να καλύπτουν την επεξεργασία του των ΑΕΕ και να αντικατοπτρίζουν το πώς έχουν σήμερα τα πράγματα. Το σύνολο των ε, προτύπων προ... και κυρίως ό,τι αφορά την επεξεργασία για νέα χρησιμοποίηση είναι κάτι που ετοιμάζουμε και θα δημοσιευθούν όσο το τέλος της φετινής χρονιάς. Ήδη κάποια πρότυπα έχουν δημοσιοποιηθεί και εδώ συμπεριλαμβάνονται γενικές αρχές για την διαχείριση των γουί, αλλά και για το τι κάνουμε με τους λαμπτήρες, με τους, ε, με τους επίπεδους πίνακες φωτισμού, καθώς και τους κυλινδρικούς ε, λαμπτήρες. Ε, θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με την ε, περισυλλογή των ε, προϊόντων σε το τέλος κύκλου ζωής που μπορεί να περιέχουν συστατικά ανθράκων. Θα φροντίσουμε να υπάρξουν τα ανάλογα πρότυπα λοιπόν για τη διαχείριση και την ανακύκλωση των ΑΕΕ και θα φροντίσουμε να υπάρξει αναγνώριση της αντιστοιχίας τους ώστε να εφαρμοστούν παρομοίως σε όλες τις χώρες. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα στην ε, παρέμβασή μου, αλλά εν τιμή ήταν σε ερωτηματολόγιο η ερώτησή σας, η προφορική ερώτηση, παρά μια απλή προφορική ερώτηση και έκανα ό,τι μπορούσα για να απαντήσω στα υποερωτήματα και όπως προείπα ελπίζω ότι δεν άφησα τίποτε αναπάντητο ή έστω κάποιο ειδικότερο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, συνάδελφε. Ο Καλ ασφαλώ. ασφαλώς. Και ευχαριστώ για τις ε, διεξοδικές απαντήσεις. Για τα κράτη-μέλη έχω μια ερώτηση. Λέτε ότι είναι πολύ διαφορετικά. Βλέπετε όμως κάποια κράτη να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα με μεγαλύτερη προσπάθεια και κάποια άλλα να μένουν πολύ πίσω, να είναι πιο αδύναμοι μαθητές. Βλέπετε κάποια κράτη που φερειπίν έχουν μεγάλους λιμένες και ευχέρεια εξαγωγών. Και όταν λέτε χρειάζονται περισσότερη έλεγχη, το αντιλαμβάνομαι, αλλά σε ποιο στάδιο θέλετε να γίνονται οι έλεγχοι. Πρέπει δηλαδή να δοθούν κίνητρα στα ίδια τα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε, σε τακτικότερους ελέγχους ή η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει αυτούς τους ελέγχους. Ποιος θα ελέγχει καλύτερα. Και το τριπλοετή ρόλο μπορεί να διαδραματίσει στην κυκλική οικονομία. Το έχουμε συζητήσει βέβαια, αλλά θα είναι ρόλος ε, ε, μοχλού, ε, θα προωθεί δηλαδή την οικονομία. Πώς θα γίνει, πώς το βλέπετε. Κύριε Σίχαουτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα και εγώ να ευχαριστήσω όπως του Καρλ για την πολύ δεξιοδική, περιστατωμένη, πλήρη απάντηση στα ερωτήματά μας. Ευχαριστούμε που θερμά. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα αισθήματα που συζητούμε εδώ, δηλαδή τη νομική αντιμετώπιση των αποβλήτων. Ένα πρόβλημα που δεν είναι καινούριο. Αντίθετος, δείχνει η μελέτη, κάτι διαφορετικό δείχνει ότι είναι διαφορετικό το φάσμα από ό,τι γνωρίζαμε, αλλά το πρόβλημα το γνωρίζαμε από πριν. Και η Επιτροπή φαντάζομαι ότι από ό,τι λέει έχει στόχο να μην χρειάζεται να ξαναγίνει ε, σε τρία χρόνια όλη αυτή η συζήτηση για την νομική διάσταση της διαχείρισης. Ζητήματα άλλα μπορεί να μείνουν. Και από τις απαντήσεις σας μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά να μην ξαναγίνει η συζήτηση η βασική για την νομική μεταχείριση. Θα είναι πολύ κακό αυτό. Πιο συγκεκριμένο τώρα, όπω λέτε και στην απάντησή σα, έχει κρίσιμη σημασία για την κυκλική οικονομία το θέμα αυτό. Στι 2 Δεκεμβρίου θα διατυπωθεί νέα ε, πρόταση για την κυκλική οικονομία. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα σε ποια ζητήματα της κυκλικής οικονομίας θα δραστηριοποιηθείτε για να δώσετε απαντήσεις. Μην μου πείτε τι έχετε ήδη ξεκινήσει, αλλά κάτι καινούριο που θα μπορούσαμε να περιμένουμε σε σχέση με την κυκλική οικονομία σε πιο ξεκάθαρους όρους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι. Ε, λοιπόν, έχετε το λόγο. Κύριε Φλόραντς, για την ερώτηση σας που νομίζω ότι αφορούσε τις εξαγωγές ή καλύτερα τις παράνομες εξαγωγές ε, α ή τα, ή τα ε απόβλητα ή απόβλητων ειδών δηλαδή και ηλεκτρονικού εξοπλισμού παράνομες. Κοιτάξτε, έχουμε έρευνες οι οποίες δείχνουν και δεν μας ξεφνιάζουν ότι τα κύρια είδη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που βγαίνουν από την Ένωση είναι τα πίπεδα. Και εκεί πέρα χρειάζεται η συμμόρφωση και οι προσπάθειες για επιβολή του νόμου. για τα ποσοστά ανακύκλησης και το μείγμα αυτής έχουμε διαφορετικές επιδόσεις των κρατών μελών και όπως είπα και νωρίτερα στην πρωτοβουλία προώθησης της συμμόρφωσης που θα ξεκινήσουμε του χρόνου. Ιδιαιτέρως θα εστιάσουμε στα κενά για τα κρατημέλη με τις χαμηλότερες επιδόσεις. συμμόρφωσης, κάτι που δεν είναι καινούριο. Ήδη γίνεται μια πρωτοβουλία προαγωγής της ε, συμμόρφωσης για τα δημοτικά απόβλητα, μια αντίστοιχη για τα επικίνδυνα απόβλητα για τα απόβλητα από οικοδομές, για πρωτοβουλία σχετική με τα οχήματα στο τέλος ζωής, όπου έχουμε πρόβλημα με τα ELVs, οχήματα άγνωστης ε, τοποθεσίας που δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται και έτσι κοιτάμε να έχουμε ένα εργαλείο που θα μας επιτρέπει πρώτα να ε, διαγιγνώσκουμε το κενό εφαρμογής και δεύτερον να εντοπίσουμε λύσεις με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των αποβλήτων. Για τη δεύτερη ερώτηση. μπορούμε. Και επικεντρώνουμε τις προσπαθίες μας στη βελτίωση της υλοποίησης χωρίς να μπορούμε να προσφέρουμε 100% ε, ε, βεβαιότητα ότι θα υλοποιηθούν και θα εφαρμόζονται πλήρως τα πάντα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αλλά πάντως είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε σημαντικές πρόοδους στα επόμενα τρία χρόνια. για τα ΑΕΕ και την κυκλική οικονομία. Δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο σε σχέση με τις επιμέρους προτάσεις. Ωστόσο η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης για την κυκλική οικονομία θα κάνει προτάσεις για τις οποίες μπορώ κυρίως να πω ή μόνο να πω ότι θα προτείνουν μέτρα που θα καλύπτουν αυτό που ονομάζεται έτερον ίμιση του κύκλου ζωής του οχήματος για ηλεκτρικό και ε, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα αποβλητά του για θέματα ε, επισκευασιμότητας, ε, διάρκεια ζωής, ανθεκτικότητας, δηλαδή πολύ σημαντικές πτυχές που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρικό ε, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και προτάσεις για την ε, ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά ώστε, και αυτό έχει τεράστια σημασία, για να δοθούν κίνητρα στη συλλογή και ανακύκλωση των ΑΕΕ. Και εν τέλει ενδέχεται και να συμπεριληφθεί στην πρόταση, την νομοθετική που θα καταθέσουμε, ε, μια ομάδα ελέγχων προδιαγραφών για ε, μηχανισμούς ευθύνης του κατασκευαστή που βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία για την διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιασμένοι για να εξασφαλίσουν τη διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων μηχανισμοί που δεν λειτουργούν σωστά. Άρα ναι, μέσω της δέσμης ε, μέτρων για την κυκλική οικονομία και χωρίς να είμαι σε θέση να δώσω πολύ συγκεκριμένε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή ως προς το περιεχόμενο των μέτρων που θα προταθούν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα προβλέπετε θετική απήχηση στη διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όχι μόνο ε, σε ύστερο στάδιο αλλά και προληπτικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτού του σημείου τη σημερινή διάταξη και να πάμε στο επόμενο. Προφορική ερώτηση για τι σπάνιε μορφέ καρκίνου και ανταλλαγή απόψεων με του εκπροσώπου τη Επιτροπή. Δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο, την κυρία Σάρμπου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Κάθε χρόνο 540.000 Ευρωπαίοι πολίτες διαγνώσκονται με μια σπάνια μορφή καρκίνου και ο όρος σπάνιος δεν χρησιμοποιείται σωστά, διότι αυτού του είδους τα καρκι... η καρκίνοι δεν είναι πλέον τόσο σπάνιοι. Είναι το 22% των νέων κρουσμάτων καρκίνου στην Ευρώπη. Το ποσοστό επιβίωσης μετά από 5 χρόνια είναι μικρότερο για όσους έχουν πληγεί από σπάνια μορφή καρκίνου σε σχέση με τους ε, ασθενεί που υπάρχουν από τι συχνέ μορφές καρκίνου. Οι πιθανότητες να μην επιβιώσουν είναι 80 έω 90% παραπάνω από όσους ε, έχουν ε, πληγεί από καρκίνο πιο συνηθισμένο όπως του ορθού ή Ε, ή άλλες μορφές. Οι περισσότεροι ε, Ευρωπαίοι πεθαίνουν από αυτού του είδους ε, τις μορφές διότι η διάγνωση γίνεται σε πολύ καθυστερημένο στάδιο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει καλύτερη ευθυγραμμισμό τη παροχή υπηρεσιών που θα συνδύζει με τι αυτές αυτέ μορφέ. Στην Ανατολική Ευρώπη το ποσοστό επιβίωσης είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη που φτάνει τα 40%. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν μια θλιβερή πραγματικότητα. Είναι σαφές ότι αν υπήρχε έγκαιρη διάγνωση αυτών των μορφών καρκίνου, εάν υπήρχε η κατάλληλη υγειονομική υπερίθαλψη, το ποσοστό επιβίωσης θα έφτανε το 80-90%. Οι έγκαιροι λοιπόν, ε, γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει παροχή υπηρεσιών και έγκαιρη πρόσβαση σε επαρκή κέντρα, σε κέντρα διάγνωσης. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή σκοπεύει να προβλέψει ελάχιστα πρότυπα για τους καρκινοπαθείς που έχουν πληγεί από αυτές τις μορφές ή και άλλες πιο συνηθισμένες και πώς προτίθεται να οργανώσει πρόσβαση σε κέντρα αναφοράς και συνεργατικά δίκτυα με διστημονική υψηλή εξειδίκευση. Ήθελα λοιπόν να θέσω εδώ τι συγκεκριμένες με ερωτήσεις. Τι δράσεις θα λάβει, αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει τα κάτω μέλη στη λήψη μέτρων ώστε να υπάρχει άγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, καθώ και μέτρα πρόληψη για του ασθενεί που πάσχουν από σπάνιε μορφέ καρκίνου, ιδίω για εκείνε τι σπάνιε μορφέ, όπου η επιστήμη μπορεί να δώσει πολύ αποτελεσματικέ θεραπείε αλλά όπου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές υπηρεσιών υγείας. Επίσης, πώς προτίθεται η Επιτροπή να παρακολουθήσει τα πορίσματα των ε, προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε ελάχιστε υποχρεωτικέ προδιαγραφέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για του ασθενεί που πάσχουν από σπάνιε μορφέ καρκίνου. Πώ θα παρακολουθεί η Επιτροπή την εφαρμογή των υπηρεσιών αυτών και τον αντίκτυπό του στου ασθενεί. Thank you, And now, from the Commission side, Mr. Michael Ευχαριστούμε την κυρία Σάρμπο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Χιούμπερ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση που αφορά μορφές καρκίνου, έναν τομέα που μας απασχολεί πάρα πολύ στα πλαίσια της καταπολέμησης του καρκίνου γενικότερα και όλων των χρόνων παθήσεων. Τώρα, θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε και ποια είναι τα στοιχεία για τους σπάνιους καρκίνους έτσι ώστε να τους ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους. Γνωρίζουμε από μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν και από την ε, σχέση μας και τις επαφές που έχουμε τα κράτη-μέλη για την πολιτική που ακολουθούν για τις σπάνιες παθήσεις και τους σπάνιους καρκίνους, πως τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν με τη χρονική στιγμή της διάγνωσης, με την πρόσβαση σε ε, θεραπείες, με τις κλινικές δοκιμές, με το μικρό αριθμό ασθενών, με την πρόσβαση σε εξειδικευμένα φάρμακα, όπως επίσης και με τις ε, βάσεις ιστών, όπως επίσης και με τα μητρώα ασθενών. Ξέρετε πως ε, είναι οι διαφορετικές παθήσεις αυτή η σπάνη ε, καρκίνη ε, στην αντιμετώπιση που τη στα διάφορα κράτη-μέλη και υπάρχουν και μεγάλες διαφορές από κράτος σε κράτος. Για το θέμα της πρόληψης δεν έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση για την πρόληψη αυτών των σπανίων καρκίνων, αλλά γενικά στον ευρωπαϊκά στον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του καρκίνου, νομίζω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ. Για παράδειγμα, τους καρκίνους που αναφέρατε εσείς στην προσωπική σας ε, ερώτηση. Υπάρχουν τα σημεία της έκθεσης στον ήλιο, της οδοντικής υγιεινής, ε, της κατανάλωσης, ε, υνοπνεύματος του καπνίσματος, της παρουσίας του μεγαλοϊού στηρίζουμε τα κράτη-μέλη στην προσπάθεια που κάνουν να είναι πιο ποδοτικό το σύστημα υγείας που έχουν με διαφορετικά μέσα και πιο συγκεκριμένα νομίζω το πώς θα εφαρμόσουν την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών στην διασυνοριακή παροχή ε, υπηρεσιών υγείας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία πρώτη πρόταση για το διαγωνισμό που θα γίνει για τις σπάνιες ε, ασθένειες που θα καλυφθούν από δίκτυα αναφοράς, τα οποία θα λαμβάνουμε και πληροφορίες για τους σπάνιους καρκίνους. Ένας άλλος τρόπος για να έχει κανείς πρόσβαση σε αποτελεσματική θεραπεία είναι η χορήγηση αδειών ε, σε φάρμακα που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους καρκίνους και αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσω ε, της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων τον οργανισμό φαρμάκων, ε, γιατί ξέρει πως το 60% των αδειών που επισπεσμένα χωρίς έχει να κάνει με αυτούς τους καρκίνους. Για να έχουμε λοιπόν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της κατάστασης, ξεκινήσαμε ένα έργο, το οποίο αναφέρεται και εσείς στην ερώτησή σας, και κυρίως για τα δίκτυα φροντίδας για τους ε, ασθενείς σπάνιων, ε, με σπάνια νοσήματα. Εδώ έχουμε χρηματοδότηση ε, για τους δίκτες για τους σπάνιους καρκίνους, τις δυνατότητες περισσότερης ενημέρωσης, καλύτερης διάγνωσης, καλύτερης διαχείρισης και με ένα σημείο έμφασης για την παιδιατρική έρευνα παιδιατρική ογκολογία, παιδιατρική διάγνωση και θεραπεία, όλα αυτά στα πλαίσια μιας ε, μελέτης που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων έρευνας. Στη βάση αυτή θεωρούμε πως έφτασε η ώρα να ζητήσουμε να εμπλακούν με πιο διαστρωμένο τρόπο τα κράτη-μέλη και να στηρίξουν τις προσπάθειες που κάνουμε. Έχουμε στρατηγική και για τα σπάνια νοσήματα αλλά και για τους καρκίνους και να γεφυρώσουμε τις αποστάσεις μεταξύ των δύο έχουμε το πρόγραμμα εργασίας για το 2015 όπου προβλέπουμε μια νέα κοινή δράση για τους σπάνιους καρκίνους. Αυτή η κοινή δράση, όταν λέμε κοινή, είναι προσπάθειες κοινέ μεταξύ των ε, διορισμένων αρμοδίων αρχών και της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ξεκινήσουν από την αρχή, ελπίζω, τη επόμενη χρόνια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με πιο δομημένο τρόπο. Βασιζόμενοι στα συμπεράσματα και στους ε, στις παραδοχές που έχετε στη δική σας ερώτηση, γιατί νομίζω ότι εσείς εντοπίσατε κάποια από τα σημεία συμφόρης, όπως επίσης η καταχώρηση, ο συντονισμός των κατευθυντήρων γραμμών, πρόσβαση στην πληροφορία και πιο συγκεκριμένα ε, κάποιοι σπάνιοι παιδικοί καρκίνοι. Το γενικό πλαίσιο της κοινή δράσης περιγράφεται στο πρόγραμμα εργασίας για το 2015, για το χώρο της υγείας. Και η διαδικασία συζήτηση αυτού του προγράμματος θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες όπου έχουμε όλους εμπλεκόμενους, δηλαδή γορονούς που εκπροσωπούν ε, παιδιά, ασθενείς κτλ. Ε, και θα συζητήσουν πώς θα συναντήσουμε, συντονίσουμε καλύτερα τη δράση μας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ποιο θα είναι το πακέτο που θα προχωρήσει. Αυτό ίσως ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες όσο συνεχίζει αυτή η διαδικασία. Είναι πάντως ξεκάθαρο πως ε, ξεκινώντας αυτή την κοινή δράση με τα κράτη-μέλη και με το πρόγραμμα εργασίας αυτή τη στιγμή δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε με πιο σοβαρό τρόπο το θέμα. Οι σπάνιοι καρκίνοι χάνονται κάπως γιατί έχουμε τη στρατηγική για τους πιο βασικούς και γνωστούς καρκίνους αφενός και των σπανίων παθήσεων και νοσημάτων ε, αφετέρου. Θα συντονιστούμε λοιπόν. Θα λάβουμε υπόψη και το τι θα πούν οι δύο συντονιστικές ομάδες που έχουμε για το θέμα των καρκίνων τη μία και για το θέμα των σπανίων νοσημάτων την άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ας ακούσουμε τους ε, βουλευτές. Η κυρία Γκροστέτ πρώτα. Ναι, θα ήθελα και εγώ να συμμεριστώ τις ανησυχίες του συναδέλφου για τους σπάνιους καρκίνους, για τις σπάνιες μορφές καρκίνου που με απασχολούν ιδιαίτερα καρκίνος στο πάγκρεας, σπάνιες μορφές παιδικού καρκίνου επίσης. Δυστυχώς ο ασθενής υποφέρει και επειδή έχει καρκίνο, αλλά και επειδή είναι σπάνια η μορφή και είναι δύσκολο μερικέ φορές να βρούμε λύσει. Και βέβαια αυτό δυστυχώ οδηγεί και σε μεταχείριση μεταξύ των ε, ασθενών. Οι τύποι αυτή καρκίνου δυστυχώ αντιμετωπίζουν την έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς των θεσμικών οργάνων, έλλειψη έρευνας για τις σπάνιες παθολογίες, διαγνώσεις καθυστερημένες συχνά όπως είπε και η Επιτροπή και μάλιστα νωρίτερα ήμουνα σε μια ομάδα εργασία για τους ενδοκρινικούς όγκους όπου ακούστηκε πως 6 με 7 χρόνια πολλές φορές περνάνε για να δοθεί διάγνωση ότι πρόκειται για τέτοιου τύπου καρκίνο. Πράγμα το οποίο έχει τεράστιες συνέπειες γιατί αναπτύσσεται σε σημαντικές διαστάσεις αυτό η αρρώστια, ενώ θα μπορούσαν να την είχαν αντιμετωπίσει νωρίτερα, εάν είχε γίνει νωρίτερα και η διάγνωση. Επίσης, απουσία ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και ενώ υπάρχει στο κείμενο της προφορικής ερώτησης η έκκληση για καλύτερη συνεργασία, για καλύτερη παρακολούθηση, ανταλλαγή πληροφοριών και συνοδεία των ασθενών που υποφέρουν από σπάνιες μορφές καρκίνου και όπως είπε και η Επιτροπή χρειάζεται ενίσχυση της εφαρμογής των ε, δικτύων για τα κέντρα αναφοράς ε, που προβλέπει η οδηγία για την διασυνοριακή παροχή φαρμακευτική πορεία θόρυψη, οποίο είναι και η συγγήτρια. Δυστυχώ όμω πιστωνουμε διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία αρνούνται να διαθέσουν δίκτυα αναφορά, δίκτυα κέντρων αναφορά. Κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ε, εγγραφούν σε αυτήν την εφαρμογή, να μην υπακούσουν σε αυτήν την εφαρμογή της οδηγία για τη διασυνοριακή παροχή φαρμακευτική περιθαλψής που θα ήταν σωτήρια για τους ανθρώπους που πάσχουν από σπάνιε μορφές καρκίνου και θα ήθελα πραγματικά η Επιτροπή να μας πει πώς προβλέπει να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή τη οδηγία και πώς σκοπεύει να πιέσει τα κράτη-μέλη για να προχωρήσει αυτοχύτερα. Και επίσης κλινικές δοκιμές πριν από τη διάθεση στην αγορά ε, φαρμάκων γίνονται όλο και πιο δαπανηρές στην περίπτωση των σπάνιων μορφών καρκίνου, γιατί χρειάζονται όλο και πιο προσωποποιημένες ή ε, οδηγίες ε, και εφαρμογή και άρα πρέπει να βρούμε μια λύση για τις κλινικές αυτές δοκιμές με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελπίζω και, με, και βέβαια για την επικοινωνιακή πολιτική σε σχέση με τις κλινικές αυτές δοκιμές επί επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πέραν τη προφορική ερώτηση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, βρίσκονται ότι η συζήτηση για το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντική. Συμφωνούμε κι εμεί ότι πρέπει <clears throat> να το εξετάσουμε σε βάθο. Αλλά να σημειώσουμε ότι στην ερώτηση γίνεται σαφή μνήμα ε, στου καρκίνου τη κεφαλή και του τραχύλου. Ε, και διευκρινίζεται ότι είναι κάποιε φορέ θανατηφόροι, αν και αν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, μπορούν να προφευθούν ε, τα θανάσιμα αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν η ερώτηση λέει ότι η επιστήμη μπορεί να δώσει πολύ αποτελεσματικέ θεραπευτικέ αγωγέ, αλλά δεν υπάρχουν υποδομέ συνήθω λόγου χάρη, και επαναλαμβάνεται αυτό το κείμενο, καρκίνη του κεφαλής και του, τραχάλου, του τραχύλου. Αυτό έχει να κάνει με το τι εννοούμε σπάνια μορφή καρκίνου. Διότι εάν υπάρχει υποδομή για την καλύτερη αγωγή, δεν σημαίνει ότι έχουν πάντοτε όλη πρόσβαση. Η σπάνια λοιπόν μορφή καρκίνου ούτε για την επιστημονική κοινότητα είναι κάτι το σαφές αλλά πρέπει να οριστεί έστω βάσει της ως προς την έρευνα που έχει χρησιμοποιήσει ως βάση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ε, καρκίνη με ποσοστό συχνότητας και εμφάνισης των κρουσμάτων κάτω του 6%. Πολλές φορές μιλάμε ε, για τους καρκίνους της ε, κεφαλής ε, με την ε, το, του στήθους, ε, της, ε, του εντέρου και συμπεριλαμβάνονται ένα σωρό υποκατηγορίες καρκίνων σε κάθε περίπτωση. Αυτά ε, μαζί ονομάζονται συνολικά καρκίνος της κεφαλής ή του εντέρου. Οπότε την καρκίνο της κεφαλής και του λαιμού, ε, του φάριγγα. Τέλο πάντων, οι περιπτώσεις αυτές καλύπτουν τόσες πολλές υποπεριπτώσεις και είναι και γνωστά τα πρωτόκολλα θεραπείας με τεχνολογικής λύσης πέρα των ε, χειρουργικών επεμβάσεων. Οπότε, μιλάμε για παθολογίες που αν τις δούμε μεμονωμένα σε όλες τις, τις εκφάνσεις έχουμε ούτως ή άλλως μια σπάνια μορφή. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η θεραπεία είναι γνωστή και εφικτή. Το ερώτημα λοιπόν είναι θα καταβάλουμε προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε ε, νόσους που μόνο από τη σκοπιά των ορισμών έχει πρόβλημα ως προς την θεραπεία της, αλλά στην πράξη αντιμετωπίζεται σε πολύ καλό επίπεδο στα διαγνωστικά κέντρα. Ας ε, διαφυλάξουμε τους πόρους μας εδώ και να είμαστε σαφείς με το τι εννοούμε για τις σπάνιες παθολογίες. Ε, οι πόροι που φυλάσσονται πρέπει οπωσδήποτε να κατευθυνθούν σε αυτές τις παθολογίες που ανακαλύπτονται ε, και ε, δεν συναντώνται συχνά στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Χιούμπερ της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, ήταν πολύ εύστοχες. Και είναι σαφές ότι αν κοιτάξουμε τι αποφάσει που λαμβάνουν τα κράτη σε σχέση με την παροχή φαρμακευτική περίθαλψη είναι καθαρά μέσα στο πεδίο αρμοδιοτήτων του. Εμεί μόνο θα μπορούμε να δράσουμε, ενθαρρύνοντα τι χώρε να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την αντιμετώπιση των μορφών καρκίνου, μια πιο συνολική αντιμετώπιση, εξέταση διαφορών ζητημάτων σε σχέση με την ανείχνευση, συνεργασία προφανώ. πολλές φορές, ε, όπως υπόθηκε, ε, περνάει πολλούς χρόνους για να γίνουν αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών, αυτό πρέπει να βελτιωθεί, αλλά είδαμε και τη διάσκεψη στη Λισαβόνα πρόσφατα ότι υπάρχουν προσπάθειες για κινητοποίηση και διάδοση πληροφοριών για αυτό το έργο, <clears throat> το υπόβαθρο τέλο πάντων που γίνεται και μπορούμε νομίζω να κοιτάξουμε πιο λεπτομερώς τι άλλο θα μπορούμε να κάνουμε, αλλά η δουλειά προχωράει. Στα δίκτυα αναφορα, ιδιαίτερα και από πλευρά των κρατών μελών προ τι δεσμεύσει του. υπάρχει πρόοδο δηλαδή στην υπόθεση αυτή, όσο και αν δεν μπορούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να προωθήσουν δραστηριότητε Σε σχέση με την ερώτηση για, τον, για το ρόλο ζήτημα του ορισμού, είναι νομίζω αληθές ότι εργαζόμαστε με βάση ένα κατάλογο που έχει πρακτικούς ορισμούς ως σημείο αναφοράς. 168 διαφορετικά, διαφορετικές ε, ομάδες σπάνιων μορφών καρκίνου και βέβαια μια κοινή δράση που θα ακολουθήσει, που θα είναι το ποιοτικό βήμα πρόοδου, γιατί θα εξεταστεί το ζήτημα και του ορισμού και της ομαδοποίησης και απαντήσεων που θα πρέπει να δοθούν ως προτεραιότητες για να προωθηθεί η δουλειά. Και θα προχωρήσει με την με τον προσδιορισμό, με τη διευκρίνηση των ε, προτάσεων για κοινέ δράσει σιγά Ίσως η κυρία Γιούλιχερ να θέλει να δώσει πιο λεπτομέρειες απαντήσει αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Προφανώ στο θέμα των κλινικών δοκιμών είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο υλοποίηση της σχετική νομοθεσίας. Περιμένουμε να δούμε στοιχεία που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ανταλλαγή με ένα σημείο εισόδου και επιτάχυνση τουλάχιστον των διαδικασιών. Και πέραν του σημείου για τις ε, δοκιμές, για τις ειδικέ ε, δοκιμές. Έχουμε επαφές με την Υπηρεσία Φαρμακών και την Επιτροπή ώστε να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την αδειοδότηση ιατροφαρμακευτικών προϊόντων όπου υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε χωρίς ε, να περιοριστεί η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα λειτουργίας, η ε, υποδοτικότητα του προβλήματος. Και αυτό βέβαια στο πλαίσιο των ε, θεραπείων και της πρόοδου στο θέμα των θεραπείων των Ισπανικών Καγινών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την απάντηση στην ερώτηση της Αντιπρόεδρου Σάρμπου, για τις απαντήσεις σας, για τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Και πάω στο επόμενο θέμα ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Ιατρική Υπηρεσία για ένα σχέδιο ε, ερευνών για, ε, για το πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας παρέκκλησης. Και παρακαλώ τον κύριο Πέτερλε να πάρει πρώτα στο λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, χαίρομαι που βλέπω εδώ εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Μετά το εργαστήριο που οργανώσαμε τον Ιούνιο για τα θέματα τη παιδιατρικής. Ασχοληθήκαμε με την ε, ε, παροχή και την αγωγή φαρμάκων που ακόμη δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία το εργαστήριο αυτό για να δούμε τι χρειάζεται να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση. 40% των παιδιατρικών φαρμάκων έχουν να κάνουν με την ε, αντιμετώπιση παιδικών καρκίνων μεταξύ των σπάνιων ε, νόσων στην Ευρώπη. Πρέπει να βεβαιωθούμε λοιπόν ότι υπάρχουν ποιοτικά φάρμακα για τα παιδιά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστούμε. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Γιούλιχερ πάλι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει στο νομοθετικό πλαίσιο γιατί έχουμε τη ρύθμιση για τα παιδιατρικά θέματα με τον κανονισμό για φάρμακα τα οποία πρόσφατα εγκρίθηκε. Μιλάμε δηλαδή για το 1 πέμπτο του πληθυσμού μας, το 20-21% του πληθυσμού μας είναι παιδιά. Και ξέρουμε όλοι πως τα παιδιά δεν είναι απλώς μικροί ενήλικες, έχουν πολύ διαφορετικούς οργανισμούς και πολύ διαφορετικές ανάγκες. Το 2002 ξεκίνησε μια διαβούλευση με τίτλο «Καλύτερα φάρμακα για τα παιδιά». Και εκεί διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχει έρευνα για αυτή την ηλιακή κατηγορία ή τουλάχιστον που να χωρίζει τα, την έρευνα σε ηλικιακές κατηγορίες και γι' αυτό μάλλον φταίνε ε, κάποιες ε, συνήθειες που έχουμε. Για παράδειγμα, οι γιατροί χρησιμοποιούν την νοσοκομιακή τους, τους εμπειρία περισσότερο από τις μελέτες τη στιγμή της συνταχογράφησης φαρμάκων. Αυτό που κάναμε είναι να εισάγουμε νομοθεσία με πολλά καινούργια εργαλεία έτσι ώστε να έχουμε ένα σχέδιο για την έρευνα για παιδιατρικά ιατρικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση το 2013 ε, για το θέμα με τη σύσταση μιας επιστημονικής ε, επιτροπής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για να ασχολείται με το θέμα δημιουργήθηκε το πλαίσιο που θα διευκολύνει την ε, παιδιατρική έρευνα και εκεί στα προγράμματα που βρίσκονταν υποδοκιμή δόθηκε και μια προτεραιότητα ή τοποθετήθηκε και σε μια ολόκληρη κατηγορία η ανάπτυξη ε, παιδιατρικών ε, φαρμάκων. Έγινε αρκετή λοιπόν έρευνα για διάφορες ασθένειες, για παράδειγμα και για κάποια, κάποιες ογκολογικές ασθένειες δεν ξέρω αν βλέπετε το διάγραμμα στα δεξιά, αλλά το 10% των, παιδιατρικών, των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας που συμφωνήθηκε έχει, και που έτρεξε έχει να κάνει με ογκολογικά θέματα. Έχουμε πια και τον κανονισμό και αυτό μας βοήθησε στο να έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα για τα νεογνά, για παράδειγμα, που ήταν μια μάλλον παραμελημένη ηλικιακή ομάδα και θέλουμε να λαμβάνουμε στοιχεία τα οποία να κατανέμονται αναηλικιακή κατηγορία των παιδιών έτσι ώστε να έχουν και τα σωστότερα φάρμακα. Αν δείτε από το 2006 και μετά πόση πρόοδο έχουμε πετύχει θα δείτε πως έχουμε πάνω από 800 σχέδια παιδιατρικής έρευνας που έχουν συμφωνηθεί, 95 έχουν ήδη κλείσει και βλέπετε πως αυξάνεται και η ανάπτυξη των σχετικών ιατρικών ε, και φαρμακευτικών προϊόντων, κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο. Το 2014 και 2015 είδαμε αυτές οι έρευνες, τα προγράμματα παιδιατρικής έρευνας, να ολοκληρώνονται όλο και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε και αυτά αποτελέσματα με νέες εγκρίσεις για προϊόντα τα οποία είναι παιδιατρικής ε, εμβέλειας και έχουμε εγκρίνει και νέα παιδιατρικά φάρμακα βασιζόμενοι σε νέους δείκτες και είναι εντυπωσιακό ο αριθμός, είναι πάνω από 120 τα φάρμακα αυτά, όπου μιλάμε και για δοσολογία ε, για τα παιδιά, η οποία περιγράφεται με ε, πιο πετυχημένο τρόπο. Μιλάμε λοιπόν για ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, μεν, αλλά το 13, 14, 15 έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ποιο είναι λοιπόν το πεδίο τώρα της παιδιατρικής έρευνας και των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας. Το νομικό πλαίσιο βασίζεται στα ευρήματα που είχαμε ε, σε κάτι που επιβεβαίωσε και το δικαστήριο, δηλαδή ότι για να ορίσουμε το πεδίο εφαρμογή της πετριατική έρευνα θα πρέπει να ξεκινήσουμε τον εντοπισμό της ασθένειας. Έτσι το περιγράφει το νομικό πλαίσιο και αυτό αποτελεί την αφιτηρία για τις έρευνες που γίνονται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φαρμάκων έτσι ώστε να αναπτυχθούν φαρμακευτικά προϊόντα. Ξεκινάμε δηλαδή από τις ενδείξεις χρήσης για τους ενήλικες και προχωράμε προς τα κάτω. Στα σχέδια προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας μπορούμε να έχουμε παρεκκλήσεις αν τεκμηριώνεται πως αυτό δεν χρειάζεται, αν δηλαδή πρόκειται για νοσήματα τα οποία επηρεάζουν μόνο ενήλικες. Για την παιδιατρική έρευνα και τα προγράμματα που έχουν σχέση με ογκολογικά νοσήματα, να σας πω πως είναι το 10% όλων των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας. Και εδώ το πιο σημαντικό είναι το εξή. Πουθενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο κανονιστικό πλαίσιο, δεν αναγράφεται ότι οι επιχειρήσεις δεν ε, μπορούν να υποβάλουν προγράμματα παιδιτρικής έρευνας και για ογκολογικές ε, ασθένειες. Άρα λοιπόν είμαστε πάντα ε, μέσα στην εντολή που επιτρέπει σε εταιρείε να μας καταθέσουν προγράμματα παιδιατρικής έρευνας και για ογκολογικά θέματα και αυτό νομίζω έχει σκοπό να παρακινήσει τις εταιρείε αυτές να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα το συζητήσουν από την στιγμή της σύλληψής του με τον οργανισμό έτσι ώστε να δούμε αν χρειάζεται να εξετάσουν και την παιδιατρική σκοπιά. Based also on the Βασιζόμενοι βέβαια και στο μηχανισμό δράσης που έχουμε για τις ενδείξεις. Να σταματήσω εδώ. Νομίζω πως οι συνάδελφοι θα το πάνε πιο κάτω το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχουμε την εισφορά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμακού, ο κ. Γκαρσία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας. Ε, δείτε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Είναι πάρα πολύ καλή γιατί μιλούμε για την υγεία των, παιδιών. Για μερικά από τα πράγματα που συζητήθηκαν στο εργαστήριο του Ιουνίου και σας απασχόλησαν και εσάς, πώς από ρυθμιστικής πλευράς αντιμετωπίζει τον ορισμό κάποιων ε, παιδιατρικών νόσων και πώς ορίζουμε και την πρόσβαση στην παιδιατρική αγωγή. Πρώτα πρώτα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ενδείξεις σε για να καθορίσουμε το αν προκύπτει παιδιατρική ανάγκη. Ε, μετά τα εξετάζει αυτά η Παιδιατρική Επιτροπή και αυτό το βλέπουμε στο μέσο της διαφάνειας. Έπειτα έχουμε μια συζήτηση σε επίπεδο ε, Επιτροπής και η Επιτροπή αυτή κοιτάζει ποιες είναι οι συνθήκες της νόσου που επιτρέπουν βάσει των όσων προκύπτουν από του ενηλίκους να καθορίσουμε τι παιδιατρικές ανάγκε. και μετά πρέπει να υπάρξει ε, συμφωνία με τον χρηματοδότη ε, της αγωγής για ένα PIP, δηλαδή ένα πρωτόκολλο ή μια ε, εξαίρεση από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι η Παιδιατρική Επιτροπή προβλέπει μια παιδιατρική τις συγκεκριμένε προποθέσει. ετσι προ... Ε, χορηγεί μια παιδιατρικη εξελιξη η χορηγει μια εξαιρεση Πρώτα απ' όλα από το άρθρο 11 του κανονισμού προκύπτει το πρώτο σημείο. Λέει εκεί ότι πρόκειται να χορηγούνται εξαιρέσεις εκεί όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι μία νόσος ή ε, ασθένεια ε, αφορά μόνον ε, ενηλίκους. Εκεί η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να μην ζητήσει παιδιατρική εξέλιξη του φαρμάκου και να δώσει εξαίρεση, να χορηγήσει εξαίρεση. Έπειτα. Ε, νόσος, αυτό το έχουμε πάρει από τον ορισμό, από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αφορά μόνο αυτό το χώρο της νομοθεσίας, τα παιδιατρικά, αλλά και άλλους νομοθετικά, άλλα νομοθετικά πεδία και τέλος, εξίσου σημαντικό, όπως είπα προηγουμένως, η αφετηρία της όλης διαδικασίας είναι ο εντοπισμός ανάγκης για την ανάπτυξη κάποιου φαρμάκου για τους ενηλίκους, οπότε μετά βλέπουμε κατά πόσον αυτό μπορεί να ε, ισχύσει και για τα παιδιά. Εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα. Κάτι που παρουσίασα και στην προηγούμενη διαφάνεια στην ουσία. Ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Ως ενήλικες μπορεί να έχουμε ρευματοειδή που δεν υπάρχει στα παιδιά από ανεσολογικής άποψης. Μπορούμε όμως να δούμε ποια είναι η συγκεκριμένη ασθένεια που μπορεί να ε, αντιστοιχεί στην κατάσταση των παιδιών, ποια πάθηση. Ε, δηλαδή την ε, νεανική ιδεοπαθή αρθρίτιδα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει λοιπόν στη χρόνια ιδιοπάθη αρθρίτιδα που ουσιαστικά είναι ε, Παθήσει που αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ή το λύμφωμα ε, στους ενηλίκους. Μπορούμε ε, να δούμε από παιδιατρική σκοπιά κατά πόσο να αντιμετωπίσει το λύμφωμα στα παιδιά, αλλά συνήθως το νευροβλάστομα συνδέεται με, την, ε, με πάθηση παιδική εκεί. Δεν χρειάζεται να εξελιχθεί κάποιο ειδικό φάρμακο. Θα μπορούσε και ο θελός αν ήθελε μια εταιρεία να το ζητήσει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε δίνουμε την ίδια αγωγή με το λύμφωμα. Έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποιες χαμένες ευκαιρίες ενδεχομένως. Στην έκθεση της Επιτροπής ΕΝΔΙ από το εργαστήριο του Ιουνίου υπάρχει μια δήλωση που λέει ότι το θέμα δεν είναι προτιμόμενη προτιμόμενοι για την αξινόμηση των παιδικών ασθενειών, των παιδικών παθήσεων. Το θέμα είναι να δούμε που υπάρχει ανάγκη για εξέλιξη ενός φαρμάκου και να δούμε κατά πόσον κάποιες ε, παθήσεις μπορεί να καλύπτουν ταυτόχρονα και την ε, περίπτωση των ενηλίκων και των ε, παιδιών. Εκεί χρειάζεται η ανάπτυξη ενός φαρμάκου για παιδιά. Και αυτό καθορίζει το επίπεδο HLT που θα εξηγήσω στην επόμενη διαφάνεια αλλά ο προτιμόμενος όρος είναι το χαμηλότερο επίπεδο και αυτό μπορεί να έχει και αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη παιδιατρικών φαρμάκων. Βλέπετε τώρα στο, στη διαφάνεια αυτή την ταξινόμηση της μέτρα. Την χρησιμοποίησε η Επιτροπή μας βάση των όσων έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο βλέπετε διαφορετικά λύματα για τους ενηλίκους, εκεί που δεν υπάρχει η επεξήγηση παιδιατρικό, με διαφορετικούς χρηματοδότες, σπόνσορες και μετά υπάρχουν παιδιατρικές ανάγκες, τις εντοπίσαμε λόγου χάρη για συγκεκριμένες παθήσεις και βλέπουμε ότι το υψηλότερο επίπεδο είναι εκεί που υπάρχει η δυτή διάσταση και αυτά συζητάμε με τις εταιρείε. Αυτά διαπραγματευόμαστε. Υπάρχει ένας πολύ καλός μηχανισμός λοιπόν για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες. Παντώ, διαρκώς καταβάλουμε προσπάθεια κατά την υλοποίηση που μπορεί να μην ήταν τέλεια από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να γίνεται μια κριτική αναθεώρηση των ε, ε, εξαιρέσεων ανατάξη όπως ε, δημοσιεύτηκαν τελευταία φορά στις 23 Ιουλίου 2015 την τελευταία φορά προβλέφθηκε εξαιρέση για μια τάξη φαρμάκων που επιτρέπει ένα σύστημα Συζήτηση στην Επιτροπή του τι ειδικέ συνθήκες μπορεί να ε, υπάρξουν για περιτρικά φάρμακα ανάλογα με τις ενδείξει που έχουμε από του ενηλίκους. Βάσει τη εμπειρία μας, πρόσφατων δεδομένων για φάρμακα και παθήσεις και το αποτέλεσμα είναι ότι ο κατάλογος των εξαιρέσεων έχει αναθεωρηθεί με, πραγματικές, ε, με πραγματικό περιορισμό των ε, εξαιρέσεων ανατάξει. Παρόλα αυτά, Κάποιες φορές χορηγούνται εξαιρέσεις ακόμη βάσει του άρθρου 11. Βάσει αυτής της προσπάθειας έχουμε λιγότερες προϋποθέσεις για εξαιρέσεις που περιορίζονται σε φάρμακα υπό προϋποθέσεις. Τα συμπεράσματα λοιπόν και μετά να δώσω το λόγο την ευκαιρία σε όσους θέλουν να ρωτήσουν να τις θέσουν είναι ότι οι παιδιατρικές ε, παιδιατρικοί κανόνες έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή πρόοδο στον τομέα των περιτρικών φαρμάκων. Είναι επίσης σημαντικό ότι μπορούμε να πετύσουμε φάρμακα εφόσον υπάρχουν ενδείξεις σε ενηλίκους, αλλά οι εταιρείε δεν ε, προκύπτουν, ε, δεν ζητούν πάντοτε πρωτοκολλά οικειοθελώ. Η πολιτική για τους όρους υψηλής αναφοράς ε, είναι κάτι που ζητούμε με τις παιδιατρικές μας μελέτες όσο το δυνατόν περισσότερο. Είμαστε στα όρια των όσων μπορούμε να κάνουμε. Επιπλέον ε, μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερο διάλογο με τις εταιρείε και συναντιόμαστε με εκπροσώπους τους για να καταλάβουμε ποιες είναι οι δυνατότητες για τις παιδιατρικέ εξελίξεις, για να μελετήσουμε παιδιατρικά φάρμακα και συναντιόμαστε επίσης με οργανώσεις ασθενών και ομάδες επιστημόνων. Και επίση που μας ενδιαφέρει να υπάρχει ε, συντονισμένη επιστημονική συζήτηση για τις συγκεκριμένε προϋποθέσεις που καθορίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για τις εμπειρίε μα και την ιατρική πρόοδο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σου. Κύριε Μπράνον, έχει το λόγο. Και μετά κύριε Γκοστέτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκλεμιστή, συγγνώμη που δεν μπορούσα να έρθει. Έχω να πω τα εξή εκ Ευχαριστούμε την αίμα που ήρθε εδώ σήμερα για να μας μιλήσει για το σημαντικό θέμα. Πριν από 9 χρόνια υιοθετήθηκε ο κανονισμός για τα παιδιατρικά φάρμακα και βέβαια έχει πολύ μεγάλη ε, απήχηση στην ε, αντιμετώπιση των παιδιτρικών νόσων. Ένα τομέα στον οποίο δεν έχουμε σημειώσει σημαντική βελτίωση ήταν στην αντιμετώπιση των παιδικών ασθενειών. 35.000 παιδιά και έφηβοι κάθε χρόνο διακυγνώσκονται με καρκίνο στην Ευρώπη, κύριο λόγο δηλαδή του θανάτου νέων ε, και παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ υπάρχουν προσπάθειε για την αντιμετώπιση πιο αποτελεσματικά των καρκίνων ενηλίκων τα τελευταία χρόνια, αυτό δεν συμβαίνει και για του καρκίνου παιδιών. Δεν φαίνεται η παιδιατρική νομοθεσία να έχει βελτιώσει την κατάσταση. Μόνο μία νέα μονάδα ογκολογίας έχει θεσπιστεί από την ε, θέση σε ισχύ τη νομοθεσία. Ε, μπορεί να υπάρχουν εξαιρέξει από την ε, απέτηση για παρουσίαση του λεγόμενου PIP, σχεδίου δηλαδή επιβεβαίωση σε παιδιατρική χρήση. Ε, υπάρχουν ε, καρκίνοι ενηλίκων που δεν εμφανίζονται στο παιδί, αλλά και το αντίστροφο ισχύει ταυτόχρονα και γι' αυτό μπορεί να είναι χρήσιμε οι εξαιρέσει αυτές, αλλά αυτό το γεγονός δεν λαμβάνει υπόψη το μηχανισμό δράση ενό φαρμάκου που μπορεί να ε, είναι ή να μην είναι αποτελεσματικό σε παιδιατρική ασθένεια. Δεν δοκιμάζονται δηλαδή ποτέ φάρμακα για τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικά σε ένα παιδιατρικό καρτίνο. 26 φάρμακα συγκεκριμένα θα είχαν δυναμικό αντιμετώπιση παιδιατρικών καρκίνων, αλλά μόνο τα μισά από αυτά μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την παρέκκληση από την ε, δοκιμή. Ε, πρέπει λοιπόν να, εξεταστεί η πολιτική, να επανεξεταστεί η πολιτική για την εξαίρεση από την ε, παιδιατρική δοκιμή και θα πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχουν ε, συνθήκες για την ε, χρήση σε παιδιά. Ε, εάν είναι βιολογική ή γενετικού τύπου ή ανομαλία που οδηγεί στην ασθένεια, τότε θα έπρεπε να υπάρχουν προσθέρες δυνατότητες για δοκιμή σε παιδιά, ενώ θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιείται όρος ποιτη και το επίπεδο ποιτη ως με, τρόπος μέτρησης για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και όχι παλαιότερη μέθοδος. Θα ήθελα να το εξηγήσετε λοιπόν αυτό, γιατί να μην ε, αξιολογείται η βιολογική ή η γενετικη ανομαλία της, ε, ως αιτία της νόσου και όχι η τοποθεσία της στο σώμα, ώστε αν αυτό το κριτήριο δηλαδή και όχι το όργανο του σώματος προσβάλλεται, γιατί έτσι μπορούμε να βρούμε πολύ πιο κοντινό συσχετισμό μεταξύ των καρκίνων ανηλίκων και παιδιών. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή του κάθε χρόνο από καρκίνο να περιμένουν ε, κάποια αναθεώρηση στο μέλλον. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα τώρα. Ευχαριστώ και κυρία Κροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα αναλάβει την έκθεση για τον παιδιατρικό κανονισμό πριν από 9 χρόνια και οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη για, τον αποϊχό του γιατί δεν βλέπουμε τις, ε, το θετικό αντίκτυπο που περιμέναμε. Με μεγάλη δυσκολία εξάλλου τον επεξεργαστήκαμε και τον προωθήσαμε, αλλά δυστυχώ μένουν πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βέβαια σημειώνω την πρόσφατη απόφαση της υπηρεσίας να αναθεωρήσει την παρέκκληση σε σχέση, τις παρεκκλήσεις ε, σε σχέση με τις παιδιατρικές έρευνες ε, σε έναν βαθμό, αλλά αυτό είναι μόνο μια σταγόνα στον κοινωνό και δεν αρκεί. Μπορεί λοιπόν και πέραν των παρεκκλήσεων ως προς ε, την διεξαγωγή αυτών των σχεδίων παιδιατρικών ερευνών να έχει αποτελέσει μέχρι τώρα αντικείμενο καταχρήσεων και είμαι οργισμένη ως προς αυτό το θέμα γιατί και είχα μάλιστα και την ευκαιρία να το εκφράζω αυτό μέχρι τώρα. 60% των παιδιατρικών σχεδίων έρευνας συσχετίζονται με τις παρεκκλήσεις αυτές από τα πρώτα πέντε χρόνια από τη θέση της εφαρμογή του παιδιατρικού κανονισμού 26 φάρμακα που θα είχαν πιθανή χρήση στην παιδιατρική έλαβαν άδεια για ενήλικες μόνο τα μισά όμως από αυτά μπόρεσαν να πάρουν την παρέκκληση σε σχέση με το σχέδιο παιδιατρικής έρευνας και γι' αυτό μαζί με την κυρία Βίλμο ότι είχαμε αποφασίσει εξάλλου να υποβάλουμε στον Επίτροπο ε, μια επιστολή με την υποστήριξη πολλών ενώσεων ασθενών για να ζητήσουμε να τοποθετηθεί στην υπόθεση αυτή. Ξέρουμε παρόλα αυτά πως ε, μεγάλος αριθμός ε, φαρμάκων που απευθύνεται σε ενήλικες θα μπορούσε μοριακά να είναι χρήσιμο και ενεργό, να είναι χρήσιμα και ενεργά τα παιδιά, γιατί η δράση τους δεν έχει να κάνει με την ποσότητα, αλλά με την ε, χρήση τιμωριακή και άρα μπορεί να είναι ε, αποδοτικά τόσο σε ενήλικες όσο και παιδιά. Ε, με επιχείρημα ότι δεν μπορεί να είναι ενεργό παρά μόνο για ενήλικες το φάρμακο, θα πρότεινα, έχει αρνηθεί αυτή την χρήση η αίμα. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν να γίνει μια πιο ελαστική εφαρμογή των παιδιατρικών ερευνητικών σχεδίων. Είναι πολύ αυστηρές συνθήκες τώρα και δεν είναι αρκετά ελκυστικές και από την άλλη πρέπει να ασχοληθούμε και με τους μηχανισμούς δράσης των μορίων όταν κοιτάμε την πιθανολόγηση χρησιμότητας φαρμάκου σε παιδιατρική χρήση. Και έχω επίσης και ακόμη μια ερώτηση για τις ε, ταχύες διαδικασίες, fast track όπως ονομάζεται, για την παρέκκληση της παιδιατρική χρήση. Υπάρχει στις ΗΠΑ μια, ένα σύστημα που ονομάζεται Clearing Hope που επιτρέπει την ε, επιτάχυνση στις διαδικασίες αυτές και καλό θα είναι να το ε, χρησιμοποιήσουμε τον χρησμό αυτό ως πηγή έμπνευση. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, πρέπει επιτέλους να κινητοποιηθούμε ούτως ώστε η, ε, τα φάρμακα σε παιδιατρική χρήση να είναι πολύ πιο ένεργα και να δίνουν αποτελέσματα για τον καλό των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεισφορά. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, άλλα μέλη που να ζητάνε το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το, φλό, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ξεκινήσω λοιπόν να αντιδρώ στις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν. Σαν άνθρωπος, αλλά και σαν θεσμός, πρέπει να σας πω πως είναι απόλυτα κατανοητό ότι υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός γιατί είναι φυσιολογικό να βλέπει κανείς πως υπάρχουν τέτοιου παθήσεις, είτε σπάνιες είτε όχι στα παιδιά για, τα, για τις οποίες δεν έχουμε καμία ενδεδειγμένη θεραπεία. Αυτό είναι κατανοητό. Θα ήθελα να επιστρέψω στον κανονισμό και στην κυρία Γκροστέτη, η οποία γνωρίζει πόσο δύσκολο ήταν τότε να καταθέσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο κατάλληλο. Η ανάπτυξη ενός νέου φαρμακευτικού ε, προϊόντος έρχεται μετά από την ε, ε, ανεξάρτητη προσπάθεια που κάνει μια φαρμακευτική εταιρεία. Οπότε εμείς θα πρέπει αφενός να στηρίξουμε την έρευνα σε θέματα που αφορούν παιδιά αλλά να φροντίσουμε να μην καθυστερούμε και την πρόσβαση σε νέα φάρμακα των ενηλίκων. Οπότε είναι μια λεπτή ισορροπία και πρέπει να δούμε λίγο τα κίνητρα, το τρόπο με τον οποίο παρακινούμε τις ε, εταιρείε, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης προϊόντων. Σίγουρα πάντα υπάρχει ανάγκη για κίνητρα. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως πολλά από, τα, από τους παιδιατρικούς ε, καρκίνους τους θεωρούμε παράλληλα και σπάνια πάθηση. Οπότε όντως ε, ευνοούνται από αυτά τα κίνητρα που δίνουμε για τα προγράμματα παιδιατρικής έρευνας αλλά και από τα προγράμματα για τις σπάνιες ε, ασθένειες. Θεωρούμε λοιπόν και με τον τρόπο αυτό απαντώ σε μια πρόταση που έγινε πως καλό είναι να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν σε μια αναθεώρηση του κανονισμού πριν το 2007. 2017. Η έκθεση όντως θα παρουσιαστεί το 2017 και θεωρούμε πως η ανάπτυξη των φαρμακευτικών προϊόντων είναι μια μακρά διαδικασία, δυστυχώς. Τώρα, το Νοέμβριο του 2015, βλέπουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κανονισμού, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να αποκομίσουμε μια πλήρη άποψη. Άρα λοιπόν αυτό το 2017 ως ημερομηνία εμάς μας ικανοποιεί για την αναθεώρηση γιατί πιστεύουμε πως χρειάζεται να έχουμε πιο σφαιρική ενημέρωση και πιο λεπτομερή ενημέρωση πριν κλείσουμε το θέμα αυτό. Δεν πιστεύουμε πως ο κανονισμός ο παιδιατρικός δεν έχει δώσει απτά πλεονεκτήματα, το αντίθετο θα έλεγα. Θεωρούμε πως ήταν εντυπωσιακέ οι εξελίξεις από τότε που τέθηκε σε ίσχυ. Ευχαριστώ πολύ για να δώσω τώρα το λόγο και στον Οργανισμό Φαρμάκων. Να ξεκινήσω λοιπόν από την τελευταία παρατήρηση που έκανε η εκπρόσωπος Κομισιόν και εγώ. Και εγώ το στηρίζω. Πιστεύω πως ο κανονισμός είναι πολύ πετυχημένος. Αυτό το οποίο μοιραζόμαστε μαζί σας είναι ο εκνευρισμός γιατί δεν μπορούμε να πάμε και παραπάνω από τα όσα θεσπίζει ο κανονισμό. Και σε τεχνικό επίπεδο έχει πάρει μεγάλη δυσκολία. Αυτή τη στιγμή η ιατρική κοινότητα συζητά το πώς θα ορίζει οντότητε, ασθένειε, παθήσεις. Και εμείς ορίζουμε μέσω ιστοπαθολογικών και ε, άλλων παραμέτρων και όχι μέσω ε, βιολογικής ε, περιγραφής. Οπότε καταλαβαίνετε πως και για τον κανονισμό τα όσα λέμε εδώ είναι σημαντικό. Και είναι υποσυζήτηση, οπότε χαιρόμαστε που ακούμε και άλλες απόψεις. Η εφαρμογή όμως δεν μπορώ να σας πω ότι είναι ελεύθερη προβλημάτων. Right. Um... I the necessity for some further discussion. Ωραία. Χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω συζήτηση, ίσως σε κάποια άλλη ε, ευκαιρία. Ίσως βέβαια η κυρία Γκροστέτ θέλει κάτι να προσθέσει. Να είσαστε όμως σύντομοι παρακαλώ. Για δύο λεπτάκια ευχαριστώ. Θα τα πω πολύ γρήγορα. Να σας υπενθυμίσω πως είχαμε την ευκαιρία να το δηλώσουμε και το ξέρει η Κομισιόν το να περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης το 2017 είναι υπερβολικά μακριά. Το έχω πει. Κατά καιρού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το χρόνο ζωής της Επιτροπής μας και της θητείας αυτής του Κοινοβουλίου. Πάει πολύ μακριά η βαλίτσα το ότι είναι πρόημο και τα λοιπά για να λάβουμε θέση. Έχουν περάσει 9 χρόνια έχουμε κάποια απόσταση και αν μας λέτε ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, εμείς δεν έχουμε αυτή την άποψη. Και ακριβώς ίσως θα έπρεπε να επιταχύνουμε και να μην περιμένουμε το 17 για αναθεώρηση του κανονισμού. Για να γνωρίζουμε τι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε έτσι ώστε να φτάνουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τα φάρμακα στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα επανέλθει το θέμα, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και από, την, και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα σήμερα. Μπορώ λοιπόν να κηρύξω τη λύση της σημερινής συνεδρίασης. Καλό σας απόγευμα.